Good afternoon, uh, Προτείνω λοιπόν να ξεκινήσουμε συνάδελφοι και είμαι βέβαιος ότι θα έρθουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι σιγά σιγά μετά από μια εντατική πρωινή σύνοδο με ενδιαφέροντα θέματα. Έχουμε εξίσου ενδιαφέροντα και το απόγευμα με πρώτα απ' όλα τις πολιτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μετά θα έχουμε την παρουσία του Επιτρόπου Τίμερμανς και ε, τέλος ε, το σύστημα πλοήγησης και ε, Θα ξεκινήσουμε ε, με την πολιτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μετά μια παρουσίαση του ελεκτικού συνεδρίου και της ειδικής έκθεσης για το μέσο των μικρομεσαίων σε δράση. Ξεκινάμε λοιπόν με τη συζήτηση ε, και έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας την κυρία Κριστίν Σράιμπερ. Η κυρία Σράιμπερ είναι η διευθύντρια του προγράμματος COSME και της πολιτικής μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα σας υπενθυμίσω ότι αναφερόμαστε στις μικρομεσαίες σε πολλά θέματα και πάντα υπογραμμίζουμε τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όταν μιλάμε για βιομηχανική πολιτική, για το Green Deal, για την έρευνα, την καινοτομία και για πολλά άλλα θέματα, σε πολλές άλλες ευκαιρίες. Είναι η πρώτη συζήτηση για την πολιτική των μικρομεσαίων που βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υλοποιήσει την πολιτική των μικρομεσαίων σε οριζόντιο, με οριζόντιο τρόπο σε διάφορα προγράμματα και πρωτοβουλίε. Έχουμε όμω την κυρία Σράιμπερ, ελπίζουμε να μας ε, κάνει μια σαφέστατη ανασκόπηση αυτών των διαφόρων ροών και πώς, ε, ποιες ήταν οι επιτυχίες, ποια ήταν τα προβλήματα, οι προκλήσεις και ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον. Έχουμε 45 λεπτά στη διάθεσή μας, λίγο λιγότερο γιατί ξεκινήσαμε με λίγη καθυστέρηση. Ωστόσο έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε και θα προχωρήσουμε ως εξής. Πρώτα θα καλέσω την κυρία Σράιμπερ να προβεί στην ε, παρουσίασή της για 10 λεπτά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τις παρεμβάσεις σας, θα δώσουμε προτεραιότητα στους συντονιστές ή τους αναπληρωτές τους. Καλό επίσης και ενθαρρύνω ε, τα μέλη που είναι παρόντα εδώ στην αίθουσα να επιδείξουν ενδιαφέρον και να παρέμβουν σε αυτό το διάλογο. Και φυσικά στο τέλος θα ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Σράιμπερ για να απαντήσει τις ερωτήσεις σας και να καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα. Κυρία Σράιμπερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας σήμερα ως Διευθύντρια ε, της Πολιτικής ΜΜΕ στην DG Grow και στο τερέχον πλαίσιο για την μικρομεσές θα δούμε και τα προκαταρκτικά στάδια για την επικείμενη στρατηγική των ΜΜΕ που είναι σε εξέλιξη και όπως ξέρετε έχει ανακοινωθεί για τις 10 Μαρτίου. Έχετε ήδη ως Επιτροπή ή με τον Επίτροπο και στην Ολομέλη έχετε κάνει ανταλλαγή απόψεων και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτός ο συνεχής διάλογος είναι πάρα πολύ σημαντικός για μας και στην τελευταία θητεία έχουμε πετύχει πολλά μαζί και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να παρευρεθώ εδώ κυρία Φοντελάιν είπε ότι οι μικρομεσαίες επιχείρησει αποτελούν όλα τα καλά στην οικονομία μας και είναι μέρος των οικονομιών που δουλεύουν για τους ανθρώπους και το Ευρωκοινοβούλιο ήταν μια ισχυρή φωνή υπέρ των ΜΕ ε και των επιχειρηματιών και υπέρμαχος. Και οι κοινέ προσπάθειε μα νομίζω έχουν επιφέρει πολλά αποτελέσματα. Αν δούμε την υλοποίηση του προηγούμενου προγράμματος COSME, που ήταν το πρόγραμμα αναφοράς για την τελευταία περίοδο, πετύχαμε πρόσβαση στη χρηματοδότηση, κάποιους αριθμούς, πάνω από μισό εκατομμύριο μικρομεσές έχουν πάρει 30 δις ε, χρηματοδότησης. Έχουμε διάφορα ε, ε, κονδύλια που δεν θα τα είχαν πετύχει αλλιώς. Έχουμε και το δίκτυο Enterprise Europe που το έχετε υποστηρίξει, 625 κέντρα οργανώσεις που έχουν ε, βοήθησει ένα τέταρτο του εκατομμυρίου μικρομεσαίων να αυξηθούν διεθνώς. Και βέβαια συρίζουμε ανθρώπους με τη φιλοδεξία να ξεκινήσουν την επιχειρήση τους. Και θέλω να ε, τονίσω τις 10.000 νέους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus μέχρι το 2020. Και ήταν μια πρωτοβουλία που αρχικά ήταν επιλοτική από το Ευρωκοινοβούλιο είχε προέρθει και είναι υπέροχη αυτή η ιδέα γιατί ε, προήλθε από το Κοινοβούλιο και ε, εξελίχθηκε. Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε και εδώ και στην ΙΜΚΟ που έχει προσελκύσει ενδιαφέρον. Έχουμε πετύχει να μειώσουμε τις καθυστερήσεις πληρωμών ε, τις καθυστερημένες πληρωμές στις μικρομεσαίες που ήταν ένα σημαντικό θέμα το οποίο καταφέραμε να μειώσουμε κατά 10 μέρες κατά μεσόωρο. Δεν είναι Μπορεί να μην ακούγεται πολύ, αλλά είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες. Υπάρχουν προκλήσεις σε αυτή την στατική που θα αντιμετωπίσουμε. Οι δύο κυριότερες είναι τα δύο κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ. Πρώτα απ' όλα έχουμε το θέμα της μετάβασης στη, σε, σε αηφόρα μοντέλα επιχείρησης και πώς να δράξουν τα ωφέλη της ψηφοποίησης. Και ε, υπάρχει και μια άλλη πτυχή, ε, διασφαλίζονταν στην κοινωνική συνοχή έτσι ώστε να μην αποκλειστεί κανείς και να ενσωματωθούν ή ΜΕ στον κοινωνικό ιστό της Ευρώπης. Να τονίσουμε ότι παρόλο που είναι εύκολο για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη να ξεκινήσουν τις λειτουργίες τους, έχουμε ακόμη δυσκολίες και θέλουμε να διευκολύνουμε τις μικρές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν και να γίνουν παγκόσμιοι ε, καινοτόμοι φορεί. Θέλουμε να εξετάσουμε αυτά τα θέματα έτσι ώστε να ε, διασφαλίσουμε ότι αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα στις νέες στρατηγικές των ΜΜΕ. Να τονίσω επίσης ότι θα κτίσουμε πάνω στις επιτυχίες που έχουμε μέχρι τώρα. Είναι σημαντικό. Η νέα στρατηγική θα στοχεύει τις ΜΜΕ όλων των μεγεθών και όλων των μορφών και τύπων, από παραδοσιακές ε, μέχρι νεοφυείς, scale-ups, ε, όλων των τύπων και ειδών και μεγεθών, αλλά θα παραμείνουμε εστιασμένοι στις υφιστάμενες προτεραιότητές μας και θα σώσουμε, ε, δεν θα ε, απορρίψουμε αυτά που έχουμε πετύχει μέχρι στιγμής. Θα προσπαθήσουμε να γεφυρίσουμε τα κενά που έχουμε εντοπίσει στις ανάγκες των ΜΕΕ. Θα συνεργαστούμε επίσης με τους διάφορου θεσμού, τα κράτη-μέλη και τους ενδιαφέρουμενου φορεί και να τονίσω το ε, SME Envoy Network που έχει σημαντικό ρόλο. Ο Επίτροπος Μπρετών αναφέρθηκε στην Ολομέλεια ότι θα ορίσει έναν εντεταλμένο για τις μικρομεσαίες σύντομα και θα σα ασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ε, μεγάλη ορατότητα και θα είναι ένας οργανικός δεσμός ανάμεσα ε, στο νοσιακό, στο εθνικό και το περιφερειακό επίπεδο. Τώρα θα ήθελα να δω ε, λίγα θέματα που είναι σημαντικά. Πρώτον είναι η καλύτερη ρύθμιση. Όταν μιλάμε με τις έψιλο είναι το κυριότερο ζήτημα που τους απασχολεί, η ρύθμιση. Και εδώ έχουμε δει ε, ότι η Επιτροπή έχει υποσχεθεί ε, καλύτερη ρύθμιση. Ε, θέλω να τονίσω ότι δεν έχουμε να μιλάμε για απορρίθμιση, αλλά για νομοθεσία ε, με λιγότερο χρονοβόρο τρόπο, πιο μεγάλη διαφάνεια, διασφαλίζοντα στις, τα πρότυπα ε, εργασίας. Και επίσης η, η αξιολόγηση επιπτώσεων. Έχουμε δοκιμές αλλά σίγουρα θα ενισχύσουμε και θα κάνουμε αυτές τις δοκιμές πιο ε, αποτελεσματικές και αυτό είναι σημαντικό εν ώψη των μέτρων που ε, θα δείτε στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας και θα, σίγουρα θα έχετε ε, σύντομα την παρουσία του Επιτρόπου εδώ και θα υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας. Έχουμε τα βασικά εργαλεία για την καλύτερη ρύθμιση, αλλά σίγουρα μπορούμε να βελτιωθούμε στο μέλλον. Σίγουρα ε, περιμένουμε τις εισηγήσεις ε, σας σε αυτή τη στρατηγική. Να τονίσουμε επίσης την ιδέα του Once Only Digital by Default. Αυτό ε, έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να δούμε επίσης το θέμα που το ακούσαμε σε αυτήν την Επιτροπή της, του, του αντικτύπου της νομοθεσίας στην κοινότητα. Αυτό είναι η αρχή του one in, one out. Επίσης θα έχει το δικό της ρόλο. Τώρα, λίγα πράγματα για την ενιαία αγορά που είναι ο σημαντικός χώρος για τις ΜΜΕ, αλλά σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί φραγμοί ε, και αυτό δεν βοηθά τις ΜΜΕ να αυξηθούν στην ενιαία αγορά και να αναπτυχθούν. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι διευκολύνουμε ε, πρωτοβουλίες από τη βάση στην κορυφή που εσείς ε, πολλές φορές ε, μας ε, προβάλλετε όταν οι ΜΜΕ έχουν δυσκολίες διασυνοριακά και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι βελτιώνουμε τα πράγματα από τη βάση στην κοροφή και πολλές φορές επίσης τα κράτη-μέλη υπερ υλοποιούν κάποιους κανονισμούς ότι ε, υπάρχουν υπερβολικοί κανονισμοί και αυτό δυσκολεύει τη λειτουργία των ΜΜΕ. Αναφέρθηκα στις καθυστερημένες πυρομές. Είναι ακόμη ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για κάποια κράτη-μέλη. Υπάρχουν ε, βουλευτές που το γνωρίζουν αυτό το θέμα. Έχουμε κάποιους τομείς όπου έχουμε τα δύο τρίτα των τιμολογιών που πληρώνονται καθυστερημένα στι κατασκευέ, στο λιανικό εμπόριο. Θα πρέπει να εξετάσουμε αυτά τα θέματα επίσης, διότι θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι ε, είμαστε ε, στην ώρα μας στις πληρωμές μας. Σε ό,τι αφορά στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση, όπως είπα, έχουμε κάποια μέτρα ε, στα πλαίσια του προγράμματος Κόσμε και θα συνεχιστούν στα πλαίσια του δεύτερου, του, του, του, επόμενου προγράμματος που θα ακολουθήσει West EU. Θα έχουμε όλα ε, ομαδοποιημένα τα ε, χρηματοδοτικά μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στους στόχους μας. θα βεβαιωθούμε ότι ενθαρρύνουμε την αηφορία των πληρωμών, της χρηματοδότησης. Για τις μικρομεσαίες επίσης αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί επιπρόσθετο άγχος και επίσης θέλουμε και το είδατε και στις κατευθυντήρες γραμμές της Πρόεδρου Φαντερλάινεν ότι θέλουμε να διευκολύνουμε τις ΜΕ να επωφεληθούν της κεφαλαίου ε, και θέλουμε να έχουμε μια πρωτοβουλία για τα IPOs. Και για να δώσω χρόνο στις ερωτήσεις, θα ήθελα να κλείσω τονίζοντας το θέμα της διεθνοποίησης στην ενιαία αγορά και και επίσης ε, της συνεργασίας όλων των οικοσυστημάτων θα, ε, είναι πολύ σημαντικά. Θέλουμε να κάνουμε καλύτερη χρήση των διαφορών δικτύων που έχουμε. Έχουμε το δίκτυο Enterprise Europe, έχουμε τα ε, innovation hubs και θέλουμε ε, οι υπηρεσίες να είναι σημαντικές και συναφείς. Σε αυτό το πλαίσιο που συνεχώς αλλάζει έχουμε διάφορες δυσκολίες στην διαπραγματεύση των συμφωνιών και θέλουμε να διαβεβαιωθούμε ότι οι ΜΜΕ εποφελούνται των πλέον εκτιμάτων. Αυτά λοιπόν ε, σε λίγα λόγια ήταν τα κυριότερα θέματα και Τώρα είμαι έτοιμη να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ελπίζω να καταφέρω να απαντήσω κιόλας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, μας παρουσιάσετε όλα τα εργαλεία και τις πρωτοβουλίες ε, και δείξατε πάρα πολλά θέματα τα οποία συζητήσαμε, πρόσβαση στην χρηματοδότηση, μείωση της ε, γραφειοκρατίας, ε, πώς ε, μπορούμε να βελτιώσουμε τα προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς μπορούμε να ορίσουμε καλύτερα τις πολιτικές μας έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τώρα πάμε στις πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να καλέσω αδέλφους να υποβάλουν ερωτήσεις θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε με το ΕΛΚ, η κυρία Βιρκούνεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Σράιμπερ, για την ε, παρουσίαση. Νομίζω ότι θίξατε πάρα πολλά και σημαντικά θέματα στην ομιλία σας, όπως ε, καλύτεροι κανονισμοί. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο για αυτή την Επιτροπή, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πολύ συχνά η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ε, φτιάχνεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ πρέπει να είναι για τις μικρές. Είναι σημαντικό το ότι η νέα Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει συνεχίσει τη δουλειά για τι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσει. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι να δούμε πω θα εφαρμοστούν όλοι αυτοί οι κανόνε. Μιλήσατε επίση ε, για το θέμα των καθυστερημένων πληρωμών. Αυτό είναι ένα θέμα που έρχεται και επανέρχεται με τις, σε σχέση με τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Πρέπει λοιπόν ε, να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η οδηγία για τι καθυστερημένες πληρωμές να εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη. Η κλιμάκωση, και αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο πρέπει πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Σήμερα αργότερα θα μιλήσουμε περισσότερο για το πρόγραμμα Horizon. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας, το πώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα Horizon. Είναι σημαντικό να υπάρχει αυτό το εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ε, εσείς ε, στην Επιτροπή, ε, ποια είναι η αξιολόγηση που έχετε κάνει. Υπάρχουν κάποιες επιτυχημένες ιστορίες που να δείχνουν τι είδου επιχειρήσεις έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα Horizon ε, και τι είναι εκείνο που κάνει το πρόγραμμα επιτυχές. Αυτά να μοιραστούν ως ε, καλές πρακτικές ε, στην Ευρώπη. Για την ψηφιοποίηση, Δείξατε και αυτό το θέμα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις λόγω της ψηφιοποίησης έχουν τώρα ένα τελείως νέο επιχειρηματικό μοντέλο. Έχουμε όμως και πολλές παραδοσιακές μικρομεσαίες που δεν έχουν τις ε, δεξιότητες για να ανταπεξέλθουν στην ψηφιακή εποχή. Και θα ήθελα να γνωρίζω ε, κατά πόσον σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχετε εργαλεία για να ενθαρρύνετε και τις ε, παραδοσιακές μικρομεσαίες οι οποίες να μπορούν και αυτές να υποφεληθούν από την ψηφιοποίηση και να επιβιώσουν από τον ανταγωνισμό ή είναι κράτη που θα πρέπει να το λύσουν τα ε, κράτη-μέλη και να διαδώσουν τις ε, καλύτερες δυνατές ε, πρακτικές. Ευχαριστούμε την κυρία Βιρκούνεν εκ μέρους του Renew Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε Χριστίν, χαίρομαι που σε ξαναβλέπουμε. Ε, στο πρόγραμμα 2020 η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να ε, εισαγάγει μια πλατφόρμα όπου εκεί θα εξετάζεται το θέμα της απλούστευσης, ε, καλύτερη ε, νομοθέτηση. Ε, ποιο είναι το όραμα πίσω από την πλατφόρμα, μήπως μπορείτε να είστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Και η πλατφόρμα αυτή πώς θα επηρεάσει τις προτάσεις της Επιτροπής. Πώς μπορεί καλύτερα να είναι σίγουρος ότι η φωνή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όχι μόνο θα ακούγεται, αλλά θα λαμβάνεται και δράση. Επίσης, ε, αυτές οι μέρες ε, βρίθουν από την ε, τεχνητή νοημοσύνη. Μιλάμε πολύ για τις μικρομεσαίες, πώς θα υποφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Υπάρχει βέβαια η δυσκολία των νεοφιών επιχειρήσεων, των μικροεπιχειρήσεων επιχειρήσεων ε, για μεγάλα προγράμματα, ίσως ε, για κάποιες μεγαλύτερες μικρομεσαίες. Το πρόβλημα είναι ο ανασχεδιασμός ε, του επιχειρηματικού τους μοντέλου, το ανθρώπινο κεφάλαιο. Η τακτική και η πρακτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε αυτέ να επωφεληθούν πλήρως από την τεχνητή νομοσύνη και από άλλες πολιτικές. Ένα βασικό στοιχείο είναι πώς μπορεί κανείς να επιτύχει το στενό διάλογο ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα σημεία επαφής ε, και τα μελλοντικά ε, κέντρα καινοτομία. Και το τελευταίο που θέλω να πω ε, για την έκθεση Ακούσαμε ότι αυτή υπάρχει αυτή η έκθεση για τις μικρομεσαίες σε μία έρευνα που έκανε το ελεγκτικό συνέδριο ε, και η έρευνα αυτή κατέδειξε ότι το 64% των επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν πλήρως τα θέματα της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα μπορούσαν να έχουν επωφεληθεί. Το 64% είναι όμως ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Έχουμε λοιπόν όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, το COSME, το EFSI. Ε, θα μπορούσαν επιχειρήσεις να επωφεληθούν περισσότερο. Τι συγκεκριμένα βήματα μπορούν να γίνουν έτσι ώστε να αναδιαμορφωθεί η επικοινωνία. Γιατί νομίζω ότι αυτό το 64% ε, πρέπει να μας κάνει να ανησυχούμε ότι δεν υπάρχει σωστή επικοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους του ID, της ομάδας ID, σας καλωσορίζουμε, κυρία Διευθύντρια. Άκουσα τη συζήτηση ε, στην τελευταία ολομέλεια των ε, Επίτροπων Μπρετών που κατά κάποιον τρόπο μας παρουσίασε ε, ποια θα πρέπει να είναι η στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άκουσα και τη δική σας την άποψη. Αυτή τη στιγμή έχουμε διακηρύξεις αρχής και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι στις προτάσεις. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πάνω απ' όλα. Η 361 του 2003, εκεί γινόταν λόγος για την Ιταλία, πολύ σημαντική αυτή η πρόταση. Ε, συζητάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η σύσταση αυτή αφορά ε, τις ε, μικρές, τις πολύ μικρές και μετά τις μεσές, γιατί σε πάρα πολλές περιοχές υπάρχει έτσι μία σύγχυση ε, ακόμα και στις μικρές επιχειρήσεις ε, με λίγους ε, υπαλλήλους που όμως και αυτές συμβάλλουν στην οικονομία του κράτους. Γι' αυτό λοιπόν εάν ισχύει αυτή η σύσταση θα πρέπει να επανέλθουμε στον ορισμό γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο επίτροπο είπε ότι ίσω θα πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό εντεταλμένο για τι πολύ μικρέ επιχειρήσει. και ε, θα δούμε ποιο θα είναι εκείνο, ο οποίο κατά κάποιον τρόπο θα μπορέσει να έρθει σε επαφή με άλλους, ε, άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μπορούσε ίσως να προτείνω κάτι και να προτείνουμε εμεί κάτι η δουλειά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την, καθυστέρηση, για την ε, οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές είναι μια πολύ καλή οδηγία. Αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις ε, βρίσκονται σε δυσκολίες και ήταν οξυγόνο αυτό που τους προσφέρθηκε. Πάντως πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική η οδηγία αυτή. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να αναθεωρήσουμε ε, την πράξη για τις μικρές επιχειρήσεις, Small Business Act, αλλά να έχουμε και μία μελέτη για μεγαλύτερη ευελιξία, κυρίως όσον αφορά το ΦΠΑ και τα απλουστευμένα ε, φορολογικά καθεστώτα για τέτοιου είδους ε, επιχειρήσεις. Τώρα, πρόσβαση στην τραπεζική πίστη ε, και αυτό θα μπορούσε να βελτιωθεί οι επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν δάνεια για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Και ένα τελευταίο θέμα όπου πιστεύω ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας, δηλαδή να υπάρχει ένας κανόνας που θα επιτρέπει την ε, ε, προέλευση των προϊόντων και το made in. Αυτό για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι σημαντικό γιατί μην ξεχνάμε βρισκόμαστε ε, σε ένα κόσμο παγκοσμιοποιημένο και έτσι οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν με αυτές τις ρυθμίσεις να προχωρήσουν λιγάκι. Ευχαριστούμε πολύ. Ίσως να απαντήσετε σε αυτές τις ε, τρεις παρεμβάσεις και μετά θα ακούσουμε άλλες ε, δύο παρεμβάσεις και αν έχουμε χρόνο στο τέλος θα μπορείτε να λάβετε και πάλι το λόγο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ στις τρεις ερωτήσεις σας. Ε, καλύψατε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων. Κύριε Βούλκονα, να σας απαντήσω το εξής. γιατί σημείωσα κάποια από αυτά τα οποία ε, είπατε για να απαντήσω συγκεκριμένα για την ψηφιοποίηση, για παράδειγμα, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχουμε ένα πειραματικό ε, project που τρέχει στα πλαίσια του κόσμος που ε, έχουμε καλύψει το θέμα της χρηματοδότησης μικρομεσαίων που έχουν ψηφιακό σχέδιο. Αυτό δεν είναι η εταιρεία που θέλει να αγοράσει υπολογιστή, όχι. Είναι μια εταιρεία η οποία μεταμορφώνεται μέσω ψηφιοποίησης και χρειάζεται ε, δανεισμό για να τα καταφέρει. Έχουμε λοιπόν το EIF το οποίο ε, δίνει αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε ξεκινήσει με τη διαγωνιστική διαδικασία και νομίζω ότι στην πρόσκληση έχουμε ήδη, για την πρόσκληση έχουν κατατεθεί ένα-δύο προτάσεις ήδη. Αυτά για τη χρηματοδότηση και οι δυο σας κάνατε ε, ερωτήσεις που καλύπτουν την τεχνητή νοημοσύνη αλλά και κάποια πιο παραδοσιακά κομμάτια. Πιστεύω ότι η στρατηγική μας αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε καλύτερα τους παραδοσιακούς μηχανισμούς χρηματοδότησης. Και βέβαια ε, θα προτείνουμε να μεγαλώσουν, να στοχεύουν σε διαφορετικές κατηγορίες μικρομεσών επιχειρήσεων και να συνδέονται μεταξύ τους, αλλά και με το υπάρχουν ε, τις υπάρχουσες δυνατότητες σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία πάντα με τα όσα γίνονται στο δίκτυο Enterprise Europe. Αυτό με φέρει στο σημείο στο νούμερο στο οποίο έδωσε η Μαρτίνα, το 64% της χρηματοδότησης. Έχουμε διαφορετικές, πολλές διαφορετικές ε, ε, προσεγγίσεις. Καταρχήν τη θηρίδα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του Invest Europe. Ε, θα το κάνουμε αυτό και για την ε, βιομηχανία του θεάματος. Τώρα, για να ξέρει κανείς πού πρέπει να απευθύνει την αίτησή του, γιατί σε κάθε εργαλείο δεν ήταν εύκολο να εντοπίσει κάθε εταιρεία που ανήκει, θα έχουμε αυτή την ενιαία θηρίδα. Επίσης, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως τα σημεία επαφής, για παράδειγμα το Enterprise Europe, το δίκτυο αυτό, θα μπορεί να κατευθύνει τις εταιρείε τις επιχειρήσεις αυτές στην καλύτερη πηγή χρηματοδότησης, στο καλύτερο ε, καθεστώς χρηματοδότησης. Και είναι σημαντικό επίσης να σας πω πως κάνουμε πολλές προσπάθειες επικοινωνίας, δημοσίευσης και αυτό είναι ένα από τα διδάγματα από το εργαλείο της μικρομεσαίας επιχειρήσης γιατί έχουμε την ΙΑΣΜΕ που είναι η δική μας ε, υπηρεσία το γραφείο δηλαδή που είναι αρμόδιο, αλλά σίγουρα μπορούν να γίνουν περισσότερα. Μας ρωτήσατε ποια είναι τα διδάγματα από το εργαλείο για τις μικρομεσαίες και θα σας πω πως έχουμε το θέμα της συνδυασμένης χρηματοδότησης, δηλαδή κατά πόσο θα είναι μέσω μετοχικού κεφαλαίου ή μέσω επιδότησης, Αυτά θα τα δούμε και θα τα σχεδιάσουμε και στο μελλοντικό εργαλείο με περισσότερη προσοχή. Κύριε Κανούτο, για τον ορισμό του τι είναι μικρομεσαία επιχείρηση, ξέρετε κι εσείς πως έχουμε και τις μικροεπιχειρήσεις, έχουμε το γενικό ε, ορισμό για το τι είναι μικρομεσαία και συνήθως όταν το διαβάζουμε έχουμε αφενός την πίεση να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι με μέτρα για τις μικροεπιχειρήσεις και αφετέρου όσους θεωρούν ότι πρέπει να διευρύνουμε τον ορισμό και θα πρέπει μάλιστα να καλύψουμε και με κάποιο είδο ορισμό και τις μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για μας είναι οποιαδήποτε, οποιοδήποτε ορισμός ε, χρησιμοποιηθεί να εφαρμόζεται σε όσο δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. Δεν θέλουμε να νομοθετήσουμε βασιζόμενοι σε εξαιρέσεις και αποκλεισμούς που δίνονται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή μπορεί να έχει κανείς μία ρήτρα και να λέει τούτη η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα στη λογιστική, στις υποχρεώσεις λογιστικής. Αλλά το να εξαιρούμε με τον τρόπο αυτό τις μικρομεσαίες κατά τη γνώμη μας δεν έχει νόημα μια και έτσι κι με μια μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεών μα είναι μικρομεσαίε. Οπότε με τον τρόπο αυτό θα εξαιρούνταν από την νομοθεσία μα. Οπότε θα πρέπει να είναι ε, ανάλογα ε, και ε, να είναι αναλογική οποιαδήποτε νέα νομοθεσία έτσι ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες των μικρομεσαίων. Αυτά ε, θέλησα να σχολιάσω. Ελπίζω να μην ξέχασα κάτι. Αν όμως κάτι ξέχασα μπορώ να απαντήσω αφού μου το ξαναρωτήσετε. Έχω και τους συναδέλφους για τον τελευταίο γύρο, οπότε και αυτοί θα σας κάνουν κάποιες ερωτήσεις. Μπορείτε να τους απαντήσετε και να δώσετε και, κάποιες, ε, και, κάποιους, και κάποια συμπεράσματα. Ο κύριος Πίβερ, καταρχήν. Θα μιλήσω γερμανικά, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Σράιμπερ, πρέπει να σας πω ότι είμαι κατενθουσιασμένος. Ε, υπήρχαν εποχές ε, πριν από κάποια χρόνια, ε, τότε οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά 70% μίλαγαν για χρήματα, για την προαγωγή, για το κόσμο, για τα διαρθρωτικά ταμεία. Η πολιτική για τις μικρομεσαίες είχε άμεση σχέση με τα χρήματα. Σήμερα ήμουν πολύ προσεκτικός και εσείς αναφερθήκατε στα χρήματα, σημαντικό αυτό, αλλά κατά 70% μιλήσατε για το πλαίσιο προϋποθέσεις πλαίσιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σημαίνει ψηφιοποίηση, ε, δίκαιη και θεμητή πρόσβαση. Πολύ σημαντικό για μένα, για μας ε, σημαίνει ότι όποτε έχουμε νομοθετική εργασία να μπορούμε να επανεξετάζουμε τις ευαισθησίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, συνθήκες, προϋποθέσεις πλαίσιο είναι one in, one out. Ε, σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει μια οριζόντια θέση ε, ένα γραφείο ε, για ε, θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αν κατάλαβα καλά, υπάρχει τέτοιο γραφείο στον κύριο Μπρετόν. Όμως πρέπει να σα πω, εμεί δεν συμφωνούμε. Το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφορά τον πρόεδρο τη Επιτροπής και όχι έναν επίτροπο που είναι σε ανταγωνισμό με του άλλου που όλοι ασχολούνται με τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Σεύκοβιτ ή Γκάμπριελ και πολλοί άλλοι έχουν σχέση με τι μικρομεσαίε. Γι' αυτό λοιπόν εμεί θεωρούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να βρίσκονται πάνω-πάνω στην πρώτη της Επιτροπής και να είναι ένα οριζόντιο θέμα, που να εξετάζεται οριζόντια. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Και έχω και ένα ερώτημα. Μιλήσατε για επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και άκουσα ότι αυτές θα σας απασχολήσουν ιδιαίτερα. Στο μέλλον, στην Πράσινη Συμφωνία. Όταν θα έχουμε ε, μικρές ε, και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα παράγουν περίπλοκα, αλλά θα έχουν περιορισμένες ε, εκπομπές. Περίπλοκη παραγωγή, αλλά με περιορισμένες εκπομπές. Και ίσως αυτές να πρέπει να ενταχθούν στην ανταλλαγή των ποσοτήτων περιορισμών για τις εκπομπές για τις μικρομεσαίες. Μήπως μπορούμε να έχουμε κάποια εξαίρεση και ίσως και στο δίκαιο για τις ενισχύσεις να έχουμε εξαιρέσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην ανταλλαγή των ε, ποσοστώσεων ε, και ως εκ τούτου συμβάλλουν καλύτερα στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Ο κύριος Μπλος. Ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη μου ερώτηση ήταν η εξή. Κοιτάξαμε τον προτινόμενο προπολογισμό από τον Σαλ Μισελ και αυτό που είδαμε ήταν ότι πρότεινε να στηριχθεί το 1 τρίτο των προγραμμάτων μόνο από αυτά τα οποία είχε προτείνει το Κοινοβούλιο. Πώς θα το αντιμετωπίσετε λοιπόν αν αυτό επηρεάζει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και για να συνεχίσουμε στη συζήτηση για το Green Deal και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πώς θα τα συνδυάσετε μεταξύ τους, πώς θα εξασφαλίσετε πως έχουν ευκαιρίες όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πως το 99% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα σεβαστούν μέχρι το 2050 τον κλιματικό στόχο για την ε, ουδετερότητα. Πώς θα μειώσουμε τις εκπομπές του άνθρακα οι ίδιοι εμείς και οι επιχειρήσεις αυτές και παράλληλα θα χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες για να είμαστε οι πρώτοι ε, οι πρωτοπόροι σε αυτή τη νέα αγορά η οποία θα είναι ελεύθερη από άνθρακα. Έτσι ώστε de facto μέσα στα σχέδια της δικής τους βιωσιμότητας και της ενεργειακής αποδοτικότητας να σχεδιάσουν επιχειρηματικά σχέδια που ευθυγραμμίζονται με τους σφαιρικότερους στόχους της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Thank you, Chair. Η κυρία Καρβάλη, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κυρία ε, Διευθύντρια που είστε μαζί μας σήμερα. Ακούγοντα τα όσα είπαν οι συνάδελφοι από το ΕΛΚ, να σα πω πω για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει, καταρχήν έχουμε το θέμα με το πλαίσιο ε, για το οποίο δεν έχουμε κάνει πολλά σχόλια, γιατί αυτέ οι διατάξει ε, ε, που λείπουν από το πλαίσιο για την πρόσβαση στην ε, χρηματοδότηση, για το δίκαιο ανταγωνισμό. Είναι τα κομμάτια που λείπουν από την ενιαία αγορά. Ας μην είναι υπερβολικά περίπλακες λοιπόν οι νομοθετικές μας ρυθμίσεις. Και έχουμε και θέματα που δεν είναι ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αρμοδιότητα των κρατών μελών. Για παράδειγμα, ε, απονομή δικαιοσύνη και η ταχύτητα τη απονομή δικαιοσύνη. Γιατί πολλέ φορέ αυτό αποτελεί μεγάλο εμπόδιο για τι μικρομεσαίε. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, ε, για να περάσει κανεί, να περάσει μια υπόθεση ε, και να τελεσυδικήσει περνάει πάρα πολλού χρόνος και διαθεσιμότητα δεξιοτήτων που είναι σημαντικό θέμα για την Ευρώπη. Ψηφιοποίηση για παράδειγμα, τεχνητή νοημοσύνη, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανθρώπους που έχουν τα κατάλληλα προσόντα και, δεξιώσεις, και δεξιότητες και δεν είναι ε, διαθέσιμοι τον αριθμό που χρειαζόμαστε στην Ευρώπη. Αύριο θα ακούσουμε τα όσα θα πει ο Επίτροπος κ. Μπρετών. Ελπίζω να μας δώσει κάποιες ε, ε, ιδέες. Χρειάζονται μηχανικοί, χρειάζονται άνθρωποι με δεξιότητες που μπορούν ε, να εργαστούν στον κυβερνοχώρο. Ο κύριος Γεωργίου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Σράιμπερ γιατί... Ευχαριστούμε, επαναλαμβάνω, και την κυρία Σράιμπερ για να το ακούσει, καθώς μας έχει καταθέσει αξιόλογες προτάσεις θα πρέπει όμω κατά την άποψή μα αυτέ οι προτάσει και οι εξαγγελίε να γίνουν έργα, να γίνουν πράξη. Θα κάνω έναν παραλληλισμό. Εάν εγώ και ο Ιουσέιν Μπορτ ξεκινήσουμε από την ίδια αφιτερία να τρέχουμε, είναι γνωστό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό υπάρχουν χώρε, υπάρχουν κράτη, υπάρχουν περιοχέ, όπω είναι ο Ευρωπαϊκό Νότο, που έχουν αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Έτσι εγώ ερωτώ στη βάση της εξαγγελίας της κυρίας Φόντερ Λάιερ, υπάρχει πραγματική πρόθεση, υπάρχει ειλικρινής πρόθεση να γίνει ένας τέτοιος ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έτσι που να μην αποκλείονται αυτές που είναι ε, μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Υπάρχει η πρόθεση να δοθεί έναν αυξημένο κονδύλι στο κόσμο. Υπάρχει η πρόθεση να γίνουν δημόσιες επενδύσεις για να στηριχτούν αυτές οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επιπλέον υπάρχει πραγματική διάθεση να γίνει αλλαγή σε κάποια κριτήρια έτσι που να μην προαποκλείονται κάποιες μικρές επιχειρήσεις όπως στη χώρα μου όπου σας λέω καταληκτικά ότι κατά έναν 99% η οικονομία δυστρέφεται σε αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και από το 13 μέχρι σήμερα στη φάση της κρίσης δηλαδή έχουν κλείσει 15.000 τέτοιες μικρές επιχειρήσεις βλάπτοντας πάρα πολύ την οικονομική ανάπτυξή της. Ευχαριστώ. Thank you so much. Σας ευχαριστώ. Αν θέλετε να δώσετε σύνομες απαντήσεις σε αυτές τις παρεμβάσεις που ακούσατε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ομαδοποιήσω οριζόντια τα θέματα, γιατί υπάρχουν κοινά σημεία. Στο θέμα της Πράσινης Συμφωνίας και της ΜΜΕ σαφέστατα η βιωσιμότητα είναι και μια μεγάλη ευκαιρία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θέλουμε να ε, βοηθήσουμε τους ηγέτες ε, στην αηφορία να θέσουν πρότυπα ε, για το μέλλον. Άρα ε, θα δοθεί στήριξη, θα δείτε σε όλα τα προγράμματα. Αυτό ε, είναι στο επίκεντρό μα. Αλλά είναι και μεγάλη πρόκληση για πολλέ, ιδιαίτερα για παραδοσιακέ μικρομεσαίε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολλέ έχουν διπλή μετάβαση ε, υψηλό κόστο μετά την ψηφιοποίηση και το περιβαλλοντικό κόστος. Και ελπίζουμε να προτείνουμε και να διαρθωρικά να τη στηρίξουμε και η χρηματοπιστωτική μας παρέμβαση εδώ στοχεύεται. Αλλά ε, εδώ έχετε τον πρώτο, τον κύριο Τίμερμαντς μαζί σας το απόγευμα. Σίγουρα θα ε, απαντήσει και έχει σχέση, ε, τα θέματα του έχουν σχέση με τις ερωτήσεις που έχει θέσει. Νομίζω είναι σημαντικό στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας, ως Γενική Αρχή θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε μια φιλόδοξη υλοποίηση. Ε, οι μικρομεσαίες πρέπει να δράξουν τις ευκαιρίε, αλλά θα πρέπει να είναι σε θέση να συμμορφώνονται και θα πρέπει να υπάρχει ένα σωστό, μια σωστή δοκιμή των μικρομεσαίων. Μαρία Καρβάλια, στι δεξιότητε. Είναι σημαντικό αυτό φυσικά και όταν ε, ρωτούμε τις μικρομεσαίες ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, είναι η πρόσβαση στις δεξιότητες. Είναι πάνω από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ψηφιοποίηση ε, θα το συζητήσετε και αύριο με την Επιτροπό μας το θέμα της ψηφιοποίησης και να θυμίσω ότι εκτός από το πακέτο που έχουμε τις 10 Μαρτίου για τις μικρομεσαίες στο βιομηχανία και την έννοια αγορά, έχουμε μια εβδομάδα μετά νομίζω ε, ένα πακέτο για τις δεξιότητες, όπου βέβαια θα εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα εις βάθος, αλλά το γνωρίζουμε, είναι ένα βασικό σημείο αυτό, κρίσιμο, το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Και τώρα θα μιλήσω γερμανικά, γιατί και εσείς μιλήσατε γερμανικά, κύριε Πίπα, όσον αφορά τον ε, ειδικό εντεταλμένο για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, το σημαντικότερο είναι η πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να είναι πιο ορατή, να υπάρχει μια πολύ καλή σχέση ανάμεσα στην πολιτική μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το εθνικό επίπεδο. Δεν μίλησα ή δεν αποφασίζω εγώ για το ποιος θα είναι ο εντεταλμένος για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν δείτε ε, λιγάκι την επιστολή του Επιτρόπου, ε, θα δείτε ότι δικό του καθήκον είναι να ορίσει τον εντεταλμένο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τότε θα αποφασιστεί και πού θα εγκατασταθεί ο άνθρωπος αυτός. Νομίζω όμως ότι έχουμε ένα κοινό στόχο, δηλαδή αυτός ο εντεταλμένος διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και διασφαλίζει το ότι σε διάφορους τομείς όπου δραστηριοποιείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι σημαντική. Και νομίζω και ο κύριος Γεωργίου έθιξε το θέμα του ε, ένα ερώτημα τώρα κατά πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα αν δούμε λιγάκι στην Ελλάδα, λέω μιλήτρια, έχουμε αρκετές παρεμβάσεις. Ε, στην Ελλάδα τώρα έχουμε ε, αρκετούς ε, αρκετή μεγάλη βελτίωση. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε κάνει καλύτερα, αλλά κάπως θα πάνε καλύτερα μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σας είπα ότι θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας ε, τα βήματα που θα ακολουθήσουμε στο μέλλον για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια, οι στρατηγικές ε, βρίσκονται ακόμα τη γενέση τους. Ε, θα κλείσω σιγά σιγά γιατί βλέπω ότι ανεπομονείτε να περάσετε στο επόμενο θέμα. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που έχει σημασία για μας ε, είναι η στρατηγική και θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν είναι ότι μόλις ε, υιοθετήσουμε τη στρατηγική πάει τέλειωσε η δουλειά για τις μικρομεσαίες. Όχι. Πολύ σωστά είπατε, οι μικρομεσαίες θα πρέπει να είναι ε, στην αιχμή του δόρατος ε, και εμείς θα βασιζόμαστε πάντα στις δικέ σα, τι αντιδράσεις. Τι θα μας λέτε εσείς από τους επιχειρηματίες σα, από τις εκλογικέ σα περιφέρειες. Είναι μια ένα διαδικασία και μόλι εγκριθεί η στρατηγική νομίζω ότι θα μπορούμε μετά να περάσουμε σε μια επιτυχημένη εφαρμογή. Ευχαριστούμε πολύ, ε, κυρία Σράιμπερ. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Ε, σας ενθαρρύνουμε να συνεχίσετε τη δουλειά σας, πολύ καλή δουλειά που κάνετε. Και ε, θέλω να σας πω ότι θα παραμείνουμε σε επαφή και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε όλες τις καλές πρωτοβουλίες για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα θα συνεχίσουμε ε, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά θα δούμε το θέμα κάτω από το πρίσμα του ελεγκτικού συνεδρίου. Θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις ε, για το πώς μπορούν να βελτιωθούν ε, τα προγράμματα τα οποία ήδη εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Μπρένιγκ Άλεξ Μπρένιγκ Μάια είναι ο Ολλανδός, μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου και σήμερα θα μας παρουσιάσει τα βασικά πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου ε, κυρίως ε, το θέμα μικρομεσής επιχειρήσεις ε, ενδράσει ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα <clears throat> για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις και ελπίζουμε ο κ. Μπρένικμαϊρ να μας παρουσιάσει και μια αξιολόγηση για την αποτελεσματικότητα ε, των μέτρων που έχουν ληφθεί για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να βελτιωθεί αυτή η αποτελεσματικότητα στο μέλλον. Συνάδελφοι, ε, αν θέλετε να λάβετε το λόγο, ε, παρακαλώ να το δηλώσετε υψώνοντας την καρτέλα με το όνομά σας, όπως συνηθίζουμε το κάνουμε τον τελευταίο καιρό. Και θα κάνουμε το εξής. Ε, θα δώσουμε 10 λεπτά για την πρώτη παρουσίαση. Ε, μετά ε, θα έχετε τις δικές σας παρεμβάσεις, προτεραιότητα έχουν οι συντονιστές, αλλά θα μπορούν ε, όλοι οι συνάδελφοι να κάνουν ερωτήσεις σε ένα γύρο και εσείς ε, θα έχετε αρκετό χρόνο ε, για να απαντήσετε στις ερωτήσεις των συναδέλφων. Τώρα έχετε το λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την ε, ευκαιρία αυτή να παρουσιάσουμε την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Επιτροπή σας. Ο τίτλος είναι «Το εργαλείο για τις μικρομεσαίες ενδράση», το κοινοτόμο αυτό πρόγραμμα το οποίο αντιμετωπίζει προκλήσεις και το βασικό μήνυμα είναι πως είναι αποτελεσματικό το εργαλείο αυτό. Και έχουμε και διάφορες προτάσεις για να βελτιωθεί, για να προσαρμοστεί αλλά είναι αποτελεσματικό. Το εργαλείο αυτό σχετίζεται με τη λειτουργία του ε, Συμβουλίου Καινοτομίας και είχα μία λεπτομερή παρουσίαση ε, σε PowerPoint αλλά πιστεύω πως καλύτερο είναι να μην τη διαβάσω όλοι, αλλά να εστιάσω σε κάποιες κομβικές διαφάνειες και θέματα. Να σας πω καταρχήν πως στην πρώτη διαφάνεια Η ερώτηση που απαντάμε είναι για ποιο λόγο ε, κάναμε αυτό τον έλεγχο. Sorry. Να σας πω λοιπόν ποιος είναι ο αριθμός των μικρομεσαίων. Το 99% είναι, συγγνώμη, είναι το 86% της απασχόλησης στην Ευρώπη. Μετά έχω το ερωτηματολόγιο του ελέγχου Δηλαδή, στοχεύσαμε στι σωστές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, γεωγραφική κάλυψη και αριστεία και το κατά πόσο στηρίχθηκαν τα καλύτερα ε, έργα μέσω του εργαλείου αυτού. Επίσης, ποια είναι τα αποτελέσματα της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αν στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ναι ή όχι μας ε, απαντήσανε με ε, τη βοήθεια των αξιολογητών, που είναι αυτοί οι οποίοι αξιολογούν τα προγράμματα που καταθέτουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως ε, και από τις μικρομεσαίες της ίδης Λοιπόν, ναι, στην πρώτη φάση μιλάμε για το τι προσελκύει τις α, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στα ευρωπαϊκά προγράμματα, διαπιστώθηκε πως το κόστος είναι δυσανάλογο και ότι υπάρχουν επικαλύψεις με αντίστοιχα καθεστώτα ή προγράμματα σε κάποια από τα κράτη-μέλη. Δεύτερη φάση που είναι τα καινοτόμα έργα είναι αυτά αποτελεσματική στήριξη. Ναι, πραγματικά εκτιμά τη στήριξη αυτή πολύ, την εκτιμούν ιδιαίτερα όλοι οι ε, ε, εμπλεκόμενοι, ε, μοχλεύει και δίνει και... και είναι και εμβληματική η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, είναι ένας στην τρίτη φάση στην διεύρυνση των αποτελεσμάτων και το κατά πόσο ωφελούνται όλοι, ναι, στηρίζει την ανάπτυξη. με μοναδικό μειονέκτημα το ότι καθυστέρησε η κίνηση και δεν ήταν ε, σχεδιασμένη ε, στο να ανταποκριθεί στις ειδικέ ανάγκες κάθε μικρομεσαίας. Γεωγραφική κατανομή. Εδώ έχουμε την αναχώρα πληροφόρηση. Παρατηρεί κανείς λοιπόν πως στην Ευρωπή έχουμε δύο κατηγορίες ε, χωρών. Μια χαμηλότερη ομάδα και μια ε, υψηλότερη στο διάγραμμα. Ποιοι βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ποια είναι η ομάδα η οποία ωφελείται περισσότερο από αυτό το εργαλείο. στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε τα δεδομένα που βλέπετε εδώ, αλλά υπάρχουν και κάποιες μη, κάποια κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη, που μπορούν επίσης να ωφεληθούν, για παράδειγμα το Ισραήλ, που ε, προσελκύει με μεγάλη επιτυχία πόρους από το εργαλείο αυτό. Πίσω από αυτή λοιπόν την γεωγραφική κατανομή στο γράφημα είναι σημαντικό να διαπιστώσουμε ποιος είναι ο λόγος που έχουμε τέτοιες διαφορές μεταξύ κρατών μελών έτσι ώστε να καταλάβουμε τι παραπάνω πρέπει να κάνει η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί η θέση των κρατών οι οποίοι ήταν στην χαμηλότερη ομάδα. Καταρχήν, διαφορετικές εθνικές στρατηγικές. Είναι σημαντικό να υπάρχει σύνδεση μεταξύ εθνικής στρατηγικής στα κράτη-μέλη Το Ισραήλ, για παράδειγμα, είναι πολύ αποτελεσματικό. Έχουν εθνικές στρατηγικές που εστιάζουν στις μικρομεσαίε και στο εργαλείο εκεί. Τέτοια στρατηγική λοιπόν θα πρέπει να έχουν για να υπερασπιστούν την καινοτομία όλα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ε, προώθησε ε, με ιδιαίτερη θέρμη το εργαλείο αυτό, οπότε μπορεί να γίνει κάτι ακόμα στις χώρες που δεν ε, ήταν τόσο πετυχημένο και επίσης έχει να κάνει και με την στήριξη που προσέφερε ή όχι το Εθνικό Σημείο Επαφής. Και αυτό είναι σημαντικό, το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα κράτη-μέλη μπορεί να παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο στο πώς λειτουργούν όλα αυτά. Και έχω και κάποιες παρατηρήσεις που έχουν να κάνουν με τη διαδικασία επιλογής Καταρχήν υπάρχουν περιορισμένοι πόροι και περιορισμένοι πόροι για τους αξιολογητές. Οι αξιολογητές μας ε, ε, απάντησαν πως ο χρονικός περιορισμός για την επιλογή τους περιορίζει υπερβολικά και ε, μειώνει τις επιδόσεις τους. Το δεύτερο που προκύπτει, και αυτό φαίνεται στο γράφημα, είναι ο αριθμός των ε, ε προγραμμάτων και έργων που υποβάλλονται ξανά και ξανά. Δηλαδή, είναι σαν να παίζει κανείς τόμπολα και αν δεν πάρω θετική απάντηση στον πρώτο γύρο θα το κατεβάσω στο δεύτερο και αν δεν τα πάω καλά και εκεί θα το κατεβάσω και στον τρίτο γύρο. Έχουμε λοιπόν τι επαναμβαλόμενε υποβολέ που αποδυναμώνουν το σύστημα γιατί χρειάζονται πάρα πολλές προσπάθειες για να αποφασιστεί η τύχη αυτών των προτάσεων με ε, αποτελέσματα τα οποία είναι περιορισμένα. Τα συμπεράσματά μας. Καταρχήν, παρατηρούμε πως είχαμε ε, αρκετές και συχνές αλλαγές στους στόχους και στις ομάδες στόχο, κάτι το οποίο δημιουργεί αβεβαιότητα. Σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Και το είχαμε δει και στην αρχή με το Horizon 2020, ότι η βεβαιότητα είναι σημαντική για να είναι ένα πρόγραμμα αποτελεσματικό. Επίσης, σημαντικός κίνδυνος του να αποκλείεται η ιδιωτική να αποκλείονται οι ιδιωτικές επενδύσεις γιατί το εργαλείο αυτό δίνει ε, επιδοτήσεις αποκλείοντας τους ιδιώτες επενδυτές. Ε, στην τρίτη φάση ε, που είναι το coaching, η συμβουλευτική δηλαδή, είναι η τρίτη φάση που έχουμε την επιτάχυνση των χειρομετικών υπηρεσιών, ε, εδώ πολύ συχνά είχαμε καθυστερήσεις. Τώρα όμως είναι στη θέση του και λειτουργεί. Και το τελευταίο συμπέρασμα είναι ότι πολλές φορές οι ωφελούμενοι χρειάζονται επιπλέον χρηματοδότηση. Να συνεχίσω λοιπόν με τις συστάσεις μας Πρέπει να βελτιωθεί η στρατηγική για την επικοινωνία και η στήριξη των εθνικών σημείων επαφής. Να βελτιωθεί η διαδικασία επιλογής και να περιοριστούν οι επανα... υποναβολές, υποβολές με συγχωρείτε, και να βρεθεί μια λύση έτσι ώστε να ε, περιοριστούν αυτές οι, οι επαναλαμβανόμενες υποβολές και θα πρέπει να ξανασκεφτούμε την πρώτη ε, ε, φάση η οποία χρειάζεται να αναπτυχθεί μετά από τα παράπονα που μας, υπέθασαν, που μας υπέβαλαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και βέβαια θα πρέπει να ε, ξέρει περισσότερο ποιοι είναι οι η Ευρωπαϊκή Ένωση και να αυξήσει τη χρηματοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρον αυτός ο έλεγχος και πολύ επικοδομητικός. Άκουσα τα συμπεράσματα και τις συστάσεις και είναι καλοδεχούμενες θα τα λάβουμε υπόψη. Συνάδελφοι, παρακαλώ, η κυρία Βιρκούνεν. Yes, thank you. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο ε, και εσά για όλα αυτά που μα είπατε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Τα διάβασα αμέσω μόλι τα δημοσιεύσατε και ε, είχε πολύ ενδιαφέρον να δει κανεί ε, τα στατιστικά δεδομένα και τι διαφορέ που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Ποιο έχει επωφεληθεί από αυτό το εργαλείο Horizon. Εγώ έρχομαι από τη Φινλανδία και πολλέ φορέ ακούμε ότι οι δικέ μα οι μικρομεσαίε δεν ξέρουν πώ να ζητήσουν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon. Τα πήγαν όμω πάρα πάρα πολύ καλά. Ε, τώρα, το θέμα της εθνικής υποστήριξης είναι καθοριστικής ε, σημασίας. Ε, ε, όλο αυτό το σύστημα των καινοτομιών, το πώς λειτουργεί είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους γιατί σε ορισμένες χώρες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι τόσο επιτυχημένες ε, που δέχονται υποστήριξη από τις χώρες τους. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική έκθεση για εμάς ε, που προγραμματίζουμε το επόμενο πρόγραμμα Horizon. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ε, τη χρηματοδότηση θα πρέπει να την παίρνουν οι καλύτερες μικρομεσαίες, όχι μόνο εκείνες που γνωρίζουν ε, πώς να ετηθούν κονδύλια. Στη συστάση σας αναφέρεται ότι θα πρέπει να ε, εξετάσουμε διάφορα εργαλεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, μήπως μπορείτε να μας ενημερώσετε για ε, τα απορίσματά σας, δηλαδή ποια είναι τα εργαλεία εκείνα που δεν λειτουργήσαν ικανοποιητικά στην ε, χρηματοδότηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή έκθεση και θα την χρησιμοποιήσουμε όταν θα εργαστούμε στο νέο πρόγραμμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και Άλεξ, ε, χαίρομαι που ήρθε. Στα τελευταία πέντε χρόνια σε βλέπω στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Ε, χαίρομαι που είσαι εδώ. Ε, που ε, θα συζητήσουμε την έκθεση αυτήν την Επιτροπή. Νομίζω ότι το έχω ήδη πει στην προηγούμενη συζήτηση ότι το 64% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν γνωρίζουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό τρομάζει. Πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ε, στις συστάσεις σας μιλάτε για καλύτερη ή καλύτερες στρατηγικές επικοινωνίες. Νομίζω θα πρέπει από κοινού να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αναδιαμορφώσει, να αλλάξει την ε, πολιτική επικοινωνίας. Πολλές φορές ε, δεν είναι γνωστές οι ανάγκες ε, των δικαιούχων. Και πώς είναι όμως δυνατόν κάτι τέτοιο. Κάθε μέρα μιλάμε για τις μικρομεσαίες. θα έπρεπε να τις γνωρίζουμε τις ανάγκες. Κατά την άποψή σας, τι, συμβαίνει, πού μπορούμε να επιτύχουμε μια βελτίωση και βεβαίως τι μπορούμε να κάνουμε ως Επιτροπή. Κατόπιν, ε, υπογραμμίζετε στην έκθεσή σας ότι τα εθνικά σημεία επαφής και οι μικρομεσαίες θα μπορούσαν να υποφεληθούν αν υπήρχαν πιο σταθεροί δείκτες προτεραιότητας. Αυτό λέγεται κάθε φορά. Δεν υπάρχουν στην αρχή σαφείς προτεραιότητες. Αν δεν υπάρχουν σαφείς δείκτες για τις προτεραιότητες, ε, δεν μπορεί να προχωρήσει όμως κανείς ε, χωρίς ξεκάθαρες προτεραιότητες, δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι εκεί που γίνεται λόγος για προσανατολισμένη υποστήριξη ε, στις μικρομεσές. Αυτό δεν φαίνεται στην έκθεση, φαίνεται δεν υπάρχει συνέχεια. Εσείς στην έκθεση σας λέτε ότι σε αυτή τη φάση ε, προκύπτει προστιθέμενη αξία. Θα ε, ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ε, πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη τα απορίσματα. Γιατί όταν λέτε ότι ναι υπάρχει προστιθέμενη αξία αλλά δεν υπάρχει ε, αντιστοιχεία, ε, κάτι δεν πάει καλά. πώ μπορούμε αυτό να το βελτιώσουμε στο μέλλον. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε πολύ κρίσιμη στιγμή, προγραμματίζουμε τα πάντα για το μέλλον, άρα ε, κάποια μαθήματα πρέπει να εξάγουμε από αυτή την έκθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με αγωνία περιμένω την επόμενη έκθεσή σα ε, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, για την έρευνα και την καινοτομία. Είσαστε ειδικό κορυφή είσαστε σε αυτά τα θέματα και προσφέρετε ε, προστιθέμενη αξία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίαση, πάρα πολύ επίκαιρη και ε, περιεκτική. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία παρουσιάζει τα πορίσματα των ε, συστάσεων. Μη στα συμμεριζόμαστε όλα αυτά, τα βρίσκουμε και πολύ χρήσιμα, κυρίως ε, εκεί ε, όπου γίνεται λόγος για επικάλυψη δαπανών, δυσκολία να έχει κανείς πρόσβαση στα κονδύλια. Στην Ιταλία, παραδείγματο χάρη, υπάρχει το εξής. Πιστεύουμε ότι τα σημεία επαφής έχουν επανδρωθεί με υπαλλήλους που έχουν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο και γιατί, διότι ε, πρόκειται και καλούνται να εφαρμόσουν εργαλεία που δεν τα γνωρίζει κανείς καθόλου καλά. Όσον αφορά το θέμα της επικοινωνίας, συμφωνώ απόλυτα με αυτά που ελέγχθησαν. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση να υπάρχουν και κάποια στοιχεία από την Πράσινη Συμφωνία. Ε, πρέπει να διερωτηθούμε κατά πόσον οι επιχειρηματίες μπορούν ε, να συμπεριλάβουν κάποια ειδικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μετά ε, να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί πάρα πολλοί από τους περιορισμούς αναφέρονται στην Πράσινη Συμφωνία. Μία ερώτηση έχω να κάνω πώς μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική η χρηματοδότηση χωρίς να τιμωρούνται οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρές. Αν λοιπόν πραγματικά επιθυμούμε να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πιστεύω ότι εμείς ως μέλη της Επιτροπής Ήτρε πρέπει να αντισταθούμε σε ε, παρεμβάσεις ε, που ίσως να είναι περιβαλλοντικά φιλικές, αλλά τελικά ε, επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις. Τέλος, ε, όσον αφορά την ε, αξιολόγηση, εκεί νομίζω ότι κάπως παίζει ρόλο το γεωγραφικό στοιχείο. Ορισμένες χώρες τιμωρήθηκαν και θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσον είναι δυνατόν να μας σχολιάσετε όλα αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ κύριε Μπόρια. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να παρέμβει. Δεν μου φαίνεται να υπάρχει. Λοιπόν, αν έχετε την καλοσύνη να απαντήσετε στις τρεις ερωτήσεις και αν θέλετε να προσθέσετε κάτι στην παρουσίασή σας και τα κατακτη τα συμπεράσματά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Θα επιχειρήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις. Το πρώτο ζήτημα, το οποίο σχετίζεται και με τις εμπειρίες στη Φιλανδία, είναι το κατά πόσον η Φιλανδία αποτελεί υπόδειγμα και είναι αποτελεσματικό και το συμπέρασμα είναι ότι είναι αποτελεσματικό ως υπόδειγμα ε, ε αν δούμε την γεωγραφική κάλυψη του ε, μέσου των ΜΜΕ στην Ευρώπη. Και ένα σημαντικό θέμα σε σχέση με αυτό ε, και που σχετίζεται επίσης και με άλλα ερωτήματα, είναι η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των Εθνικών Κέντρων Στήριξης στο Εθνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στις συνεντεύξεις που κάναμε σε διάφορες χώρες, παρατηρήσαμε ότι, για παράδειγμα, σε ορισμένες χώρες τα προβλήματα είναι τα εξής. Οι μικρές και μεσαίες επιχείρησεις και οι επιχειρηματίες δεν εμπιστεύονται τους κυβερνητικούς θεσμούς. Και είναι ένα θέμα που κυριαρχεί ε, στις δύο ομάδες της Ευρώπης. Επίσης, είχατε θέσει μια ερώτηση σε σχέση με τα διαφορετικά χρηματοδοτικά μέσα. Η Επιτροπή μπορεί να κάνει συνέργειες με άλλα χρηματοδοτικά μέσα Κατά πρώτο λόγο, η Κομισιόν θα πρέπει να γνωρίζει τις ανάγκες των δικαιούχων. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό. Μέχρι στιγμής αυτό γινόταν σε περιορισμένο βαθμό. Δηλαδή, το ερώτημα είναι, ε, πρόκειται περί ενός δανείου και ενός κονδυλίου ή υπάρχει κάποια διαφοροποίηση στις μικρομεσαίες. Νομίζω αυτή είναι μια πρόκληση για την Κομισιόν να επισέλθει σε αυτό το διάλογο, σε αυτές τις ερωτήσεις και να εντοπίσει τις ανάγκες για στήριξη των μικρομεσαίων. Η Κομισιόν θα πρέπει να διερευνήσει ευκαιρίες συνεργασίας με εθνικά Ινστιτούτα, ε, που θα βοηθήσει την Κομισιόν να ανακαλύψει περισσότερα στοιχεία για τις ανάγκες των εθνικών μικρομεσαίων σε διάφορες χώρες ή σε διάφορες περιοχές και η Κομισιόν θα πρέπει να θεσπίσει ε, στρατηγικές επικοινωνίας και μάρκετινγκ ε, μαζί ε, με τα ευρωπαϊκά ε, προγράμματα χρηματοδότησης. Έχουμε παρατηρήσει ότι σε μερικές χώρες υπάρχει επικάλυψη ανάμεσα στο τι κάνει η Κομισιόν και στο τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να γίνουν πιο εξατομικευμένες προσπάθειες και θα είναι πιο χρήσιμο σε αυτό από αυτή την άποψη. Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία ανάμεσα ε, σε παρόχους κεφαλαίων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Μέχρι στιγμής αυτή η προσπάθεια ήταν κατακαιρματισμένη. Ε, θα πρέπει να ε, εναρμονιστούν και να ευθυγραμμιστούν οι προσπάθειες του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα. Κυρία Γιαμπάλοβα, έχετε παρατηρήσει ότι το 34% δεν γνωρίζει για αυτό το μέσο και είπατε ότι αυτό είναι φαντικό. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι κρίσιμο η γνώση το... και η ευαισθητοποίηση περί του μέσου είναι σημαντική. Ε, είχαμε πει στην Κομισιόν να αυξήσει την επικοινωνία με τον έξω κόσμο και να συμβάλλει σε αυτό, γιατί μετά από αυτή τη συνάντηση θα πάω στις, SM, στις ΜΕ της Ευρώπης και θα ε, δώσω τα ίδια μηνύματα και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να ευαισθητοποιήσουμε ε, ε της μικρομεσαίας για την ύπαρξη αυτού του μέσου. Έχω επίσης παρατηρήσει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσω των Εθνικών Σημείων Επαφής η Επιτροπή να μάθει ποιες είναι οι ανάγκες των ΜΜΕ. και πιστεύω μπορούν να βελτιώσουν τις γνώσεις τους ε, για τις ανάγκες των μικρομεσαίων. Τονίσατε τη σημασία ε, μιας ε, σταθερής τοποθέτησης προτεραιοτήτων. Πιστεύω ότι μέσα σαν κι αυτό είναι σε εξέλιξη. Η Κομισιόν κινείται βήμα-βήμα. Ε, υπάρχει η εξέλιξη του προγράμματος που είναι γίνεται αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Κομισιόν θα πρέπει να σταθεροποιήσει τους στόχους που θέτει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σχετικά με την φάση 1, έχουμε παρατηρήσει δύο ζητήματα. Κατά πρώτο λόγο, η φάση 1 είναι αποσυνδεδεμένη. Κατά δεύτερο λόγο, η εκτίμηση ενός μέσου για τη χρηματοδότηση φάσης 1 έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό το λόγο συμβουλεύουμε την Κομισιόν να επαναμελετήσει το μέσο της φάσης 1 υπό την έννοια ότι πολλές συναφείς ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν στις πρώτες ε, πρωτοβουλίες και ε, θα μπορούν να ε, ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογή του μέσου αυτού. Τέλος, κύριε Μπόρκια, θέσατε κάποια ερωτήματα για την Πράσινη Συμφωνία και εκφράσατε και τις ανησυχίες σας σχετικά με την αιρεσιμότητα και το βάρος που τίθεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυτή την αιρεσιμότητα της προϋποθέσεις. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι σε μεγάλο βαθμό υπάρχουν συνέργειες ανάμεσα στο μέσο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την Πράσινη Συμφωνία. Υπάρχουν αρκετές συνέργειες και άμα αναλύσουμε τις χορηγίες του 2018 βλέπουμε ότι 40% των επιχορηγούμενων προγραμμάτων είχαν σχέση με περιβαλλοντικά θέματα, ενέργεια, τρόφιμα και μεταφορές. Σε κάποιο βαθμό λοιπόν ε, η Κομισιόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, άλλα προγράμματα σε άλλους τομείς, όπως είναι η βιομηχανία, 4% ή το διάστημα. Επίσης μπορεί να έχουν μια συνιστόσα που να σχετίζεται με την Πράσινη Συμφωνία. Πόροι που διατίθενται μέσω της Πράσινης Συμφωνίας και ιδιαίτερα μέσω των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών σέμων μπορούν να επωφελέσουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια γραμμή ανάπτυξης προς τη σωστή κατεύθυνση. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν ότι ε, αν οι προσπάθειες ε, της Κομισιόν στην Πράσινη Συμφωνία υπονοούν ότι το διοικητικό άχθος ε, είναι υπερβολικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τότε χάνουμε τους στόχους μας σε αυτή την πρωτοβουλία. Πρόεδρε, νομίζω έχω καλύψει τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί. Μάλιστα, τις έχετε καλύψει λεπτομερέστατα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την παρουσία σας, για τις απαντήσεις, για τις συστάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές για τους θεσμούς που υλοποιούν τα προγράμματα, αλλά και πολύ συναφείς για μας που είμαστε υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής και που θα ε, εκδίδουμε συνεχώς συστάσεις έτσι ώστε να αυξήσουμε την ισχύ και την παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ε, βιομηχανία και την οικονομία της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ. Θα παραμείνουμε σε επαφή. Συνάδελφοι, πέντε λεπτά διάλειμμα προτού ε, έρθει ο Αντιπρόεδρος Τίμερμανς ενώπιν της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. AUTHORWAVE Dear colleagues, uh, I propose to start again our uh, session for today. Uh. Συνάδελφοι, ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Για πρώτη φορά νομίζω φιλοξενούμε, τουλάχιστον σε αυτή τη θητεία, ε, φιλοξενούμε τον κύριο Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος είναι εκτελεστικός αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ε, η Πράσινη Συμφωνία, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το Δεκέμβρη του 2019, είχαμε μια ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία αναφέρει τις δράσεις που πρέπει να αναπτυχθούν σε θέματα περιβάλλοντος και κλίματος. Θα έλεγα ότι είναι η πιο σημαντική μας πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε πολύ φιλόδοξους στόχους και βεβαίως δεν είναι εύκολο να εφαρμοστούν όλα αυτά. Αλλά αν τελικά εφαρμοστούν, πιστεύω ότι θα αλλάξουν ε, ριζικά οι οικονομίες, οι κοινωνίες, θα, βελτιωθούν, ε, θα βελτιωθεί ουσιαστικά το περιβάλλον. Μια μισή ώρα έχουμε στη διάθεσή μας για το θέμα αυτό. Ε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αρκετοί συνάδελφοι έχουν ήδη εγγραφεί στον κατάλογο των ερωτώντων τέσσερις γύρους παρεμβάσεων θα έχουμε, γιατί έχουμε πολλούς συναδέλφους και είμαι σίγουρος ότι θα υποβάλλετε πολλές και συγκεκριμένες ερωτήσεις και είναι σημαντικό ο Αντιπρόεδρος κ. Τίμερμανς να απαντήσει στις ερωτήσεις. Ξεκινάμε δίνοντας τον λόγο στον κ. Τίμερμανς για 10 λεπτά, μετά θα ακολουθήσουν οι συντονιστές για ερωτήσεις και θα έχουμε και ε, δύο γύρους ε, με ερωτήσεις ε, συναδέλφων. Να δώσω λοιπόν το λόγο ευθύ αμέσω στον κύριο Τίμερμανς. παρακαλώ να μας παρουσιάσετε το όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, ποιες είναι οι λεπτομέρειες που έχουν προκύψει από τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα τον τελευταίο καιρό μετά την ανακοίνωση και μετά το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Πράσινη Συμφωνία. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Είναι η πρώτη μου ευκαιρία για να συζητήσουμε για την Πράσινη Συμφωνία και ε, όλα αυτά γίνονται με τεράστια υποστήριξη της κοινή γνώμης για την Πράσινη Συμφωνία και έτσι έχουμε την ευκαιρία ε, να ε, συνδυάσουμε τις περισσότερες προκλήσεις. Βεβαίως πρώτα απ' όλα την κλιματική πρόκληση. Για δέστε τι γίνεται στον καιρό πλημμύρες σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ή στην Ισπανία ο παγετός στην Ισπανία και πολλές άλλες ε, ε θεομηνίες. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα ε, να έχουμε μια αναπτυξιακή στρατηγική την ε, εποχή της βιομηχανικής επανάστασης. Βρισκόμαστε εν μέσω μιας ε, βιομηχανικής επανάστασης που είχε καταστροφικές συνέπειες. Όμως ε, όλα αυτά προσφέρουν και ένα τεράστιο δυναμικό για μια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς, νέες θέσεις απασχόλησης, διαφορετικές θέσεις απασχόλησης. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωση. Δύσκολο αυτό. Και πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος να μείνουν πίσω μερικοί. Ε, αυτή είναι η δεύτερη πρόκληση. Η τρίτη τώρα, συγκεκριμένα για την Ευρώπη, είναι το δημογραφικό πρόβλημα. Που σημαίνει ότι πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα, να δώσουμε στους πολίτες μας τις δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι παραγωγικοί και επιτυχημένοι ε, σε μια οικονομία που προκύπτει από τη βιομηχανική επανάσταση την Πράσινη Συμφωνία τη βλέπω τη δυνατότητα της Ευρώπης να συνδυάσει αυτές τις τρεις προκλήσεις και να τις μετατρέψει σε ευκαιρίες. Εγώ θεωρώ κυρίως ε, για την Ήτρε ότι εσείς θα ενδιαφέρεστε για το μεσαίο κομμάτι, δηλαδή πώς μπορούμε να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία μας με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την ε, κλιματική κρίση και παράλληλα να προσφέρει και ευκαιρίες με βιώσιμο τρόπο. Ε, σύντομα θα εκδώσουμε ένα πρόγραμμα κυκλικής οικονομίας που είναι η συνέχεια αυτών που έχουμε ήδη κάνει. Μετά θα εστιάσουμε στο τι πρέπει να γίνει για να ε, μην ε, να σταματήσουμε να ε, σπαταλάμε προϊόντα ε, στην οικονομία μας, να μην σκάβουμε, καίμε και μετά να μην πετάμε προϊόντα, να έχουμε μια κυκλική οικονομία. Αν δεν λάβουμε δράσεις, χρήση, η χρήση των μετάλλων, τα πλαστικά θα διπλασιαστούν και μέχρι το 2050 θα πρέπει να έχουμε τρεις ε, πλανήτες ε, για να ε, μπορέσουμε να συνεχίσουμε με το ίδιο καταναλωτικό μοντέλο. Αυτό βέβαια δεν επιτρέπεται. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λέμε σε κάποιους ότι ξέρετε εσείς δεν μπορείτε να αναπτυχθείτε όπως έχουμε αναπτυχθεί, έχουμε αναπτυχθεί εμείς. Πολλοί ποτέ δεν το δεχτούν και αυτοί που δεν έχουν αναπτυχθεί είναι πολύ περισσότεροι από εμάς. Ε, γι' αυτό λοιπόν α εκμεταλλευτούμε το δυναμικό που υπάρχει. Νομίζω ότι πρέπει να αυξηθεί ε, το ποσοστό του υλικού που θα εντάσσεται στην κυκλική οικονομία. Ε, τα απορρίμματα από κόστος θα τα μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Και ε, βεβαίως ε, τίποτα δεν είναι απλά πράσινο. Το θέμα είναι να βεώσουμε τους πολίτες μας ότι θα επενδύσουμε σε μια νέα οικονομία στο κέντρο της ε, κυκλικής οικονομίας που θα παρουσιάσουμε θα είναι μια πρωτοβουλία με βιώσιμα προϊόντα και μπορώ να προβλέψω ότι αυτό θα το αλλάξει όλο το παιχνίδι γιατί η πολιτική αυτή θα ασχολείται στη μετατροπή του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης το πώς τα προϊόντα μας μπορούν να είναι βιώσιμα ε, και προσιτά παράλληλα, γιατί αυτό αξίζει στους πολίτες μας. Λάβαμε υπόψη μας τις προτάσεις του Κοινοβουλίου να επεκταθεί το έβρος του οικολογικού design, να λαμβάνουν υπόψη τα βιώσιμα προϊόντα. Δηλαδή η πολιτική μας θα είναι ευρεία, συγκεκριμένη, γιατί φοβάμαι ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για όλους μας. Πάρτε λιγάκι αυτή τη γενική υποστήριξη για την ιδέα της ε, Πράσινης Συμφωνίας. Ε, υποστήριξη όμως χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα μέτρα, γιατί ορισμένα από αυτά ε, θα δημιουργούν προβλήματα, αναταραχή οι άνθρωποι. Ε, θα πρέπει όμως να καταλάβουν και τις ευκαιρίες που θα προσφέρουν. Ε, όλα αυτά ε, νομίζω θα είναι ευχάριστα για τους πολίτες όταν τα προϊόντα θα διαρκούν περισσότερο, θα χρησιμοποιούμε περισσότερα ανακυκλώσιμα υλικά και ε, τα προϊόντα να μην καταστρέφονται πριν λήξει διάρκεια της ζωής τους. Αυτή η πολιτική σημαίνει ότι θα ζητάμε από τους καταναλωτές να επισκευάζουν τα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν Νομίζω λοιπόν ε, αυτά όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Για σκεφτείτε, ε, να επισκευάζουμε ε, τα κινητά μας τηλέφωνα πριν τα πετάξουμε. Νομίζω ότι αυτές οι δράσεις μπορούν να βοηθήσουν τους πολίτες που ενδεχομένως ανησυχούν ότι δεν μπορούν να αγοράσουν βιώσιμα προϊόντα, ε, που ανησυχούν γιατί δεν θέλουν να σκεφτούν το ε, τέλος του πλανήτη. Πολλοί δεν σκέφτονται, δεν έχουν τέτοιες γιατί ανησυχούν για το τέλος του μήνα, πώς θα τη βγάλουν μέχρι το τέλος του μήνα. Γι' αυτό λοιπόν η οικονομία να δουλέψει για τους ανθρώπους. Η πολιτική μας η βιώσιμη θα καθοριστεί μαζί με την βιομηχανία. Ε, εμείς έχουμε ουσιαστικά ουσιαστικά πρότυπα, πρότυπα για λιγότερη ενέργεια να μειωθεί, το αποτύπωμα του άνθρακα, ε, να είμαστε όλοι σίγουροι ότι ε, δεν θα καταστραφεί ε, το αποθεματικό μας των υλικών. Μπορούμε να ξεκινήσουμε ε, σε τομείς όπως είναι η επικοινωνία, οι μπαταρίες, τα υφάσματα, ε, οι συσκευασίες και μετά να αναπτύξουμε περισσότερο την οικονομία μας. Όπως γνωρίζετε, με το πρόγραμμα δράσης για την κυκλική οικονομία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιό της για μια βιομηχανική πολιτική ε, σε τέσσερις φάσεις. Θα προσφέρουμε υποστήριξη στις αλυσίδες βιομηχανικής αξίας που είναι στρατηγική σημασία για το μέλλον μας. Για μένα αυτές είναι οι αλυσίδες αξίας ε, που είναι και βιώσιμες, ε, καθαρή κινητικότητα, καθαρός χάλιβας, ε, υδρογόνο, μπαταρίες για την ηλεκτρική κινητικότητα και ακόμα και με αυτές τις αλυσίδες η καλύτερη επιλογή είναι να είμαστε κυκλικοί παράδειγμα. Αν μπορούμε να κυκλώσουμε τις μπαταρίες μας με βιώσιμο τρόπο μπορούμε να στηρίξουμε σημαντικά τα καθαρά αυτοκίνητα του μέλλοντος. Και αν αυτές οι μπαταρίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκίνητα θα υπάρξουν άλλες εφαρμογές, ξέρω πολλές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μοιάζουν πολύ ελπιδοφόρες. Σήμερα θέλω να καλέσω αυτή την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν το τεράστιο δυναμικό, ε, τα προγράμματα κυκλικής οικονομίας ε, μπορούν να αποτελέσουν τμήμα των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα. Και υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες για την βιομηχανία. Ε, να εκφράσω την εξή σκέψη. Για να λειτουργήσουν όλα αυτά πρέπει όλοι να μας στηρίξουν, όλοι να συμμετέχουν. Η κοινή γνώμη, η βιομηχανία, η ακαδημαϊκή, ε, τα μέσα ενημέρωσης και ε, όσοι χαράσουν πολιτική, όλοι ε, βρίσκονται στην ίδια ε, πλευρά. Κανείς δεν πρέπει να μείνει καθυστερημένα πίσω. Ε, πάντα ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις ε, για να μπορείτε κι εσείς να αποφασίσετε ε, τι θα γίνει στους διάφορους τομείς. Και πραγματικά θέλω να ακούσω τις απόψεις σας σε όλα αυτά. Ένα σημαντικό στοιχείο θα είναι η μετάβαση, η ενεργειακή μετάβαση. Η ενεργειακή μετάβαση είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι καθοριστική σημασίας για να επιτύχει η Πράσινη Συμφωνία. Ε, πρέπει να έχουμε ανεξαρτησία από τα ορυκτά καύσιμα και να διασφαλίσουμε ικανοποιητικούς ενεργειακούς πόρους για να τρέξει η οικονομία μας και στο μέλλον. Και αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστούμε πολύ περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από αυτή που έχουμε σήμερα. Βιώσιμη ενέργεια, αιωλική ενέργεια. Αυτό ε, σημαίνει και βλέπουμε ότι προχωράει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε. Αλλά πολύ συχνά λείπουν οι υποδομές, ε, τα δίκτυα για να μεταφερθεί η ενέργεια εκεί που πρέπει και σίγουρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε την ενέργεια όταν την παράγουμε και να την χρησιμοποιούμε όταν τη χρειαζόμαστε. Αυτά είναι τεράστια έργα, επ' αυτών πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις για να υπάρξει και μετάβαση. Ε, Χωρίς το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να γίνει τίποτα και γι' αυτό τελειώνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω για το ψήφισμα γιατί αυτή είναι η μεγαλύτερη υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας μέχρι σήμερα. Και έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι ακολουθούμε την ίδια πορεία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Εκτελεστική Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για τα όσα είπατε και είναι σημαντικό το θα πρέπει να συνεργαζόμαστε έτσι ώστε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο να πετύχει. Τουλάχιστον αν δεν πετύχουμε την ομοφωνία να έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό δυνατών ε, ανθρώπων που θα συνεργαστούν για να προχωρήσουμε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σας στηρίζουμε ευρύτατα. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιες είναι οι λεπτομέρειες και λείπουν οι πλειοψηφίε στα συγκεκριμένα και θα το καταλάβετε αυτό με τι ερωτήσεις των συναδέλφων που θα είναι σίγουρα πολύ συγκεκριμένες. Να δώσω λοιπόν κατευθείαν το λόγο στους συντονιστέ, τρία λεπτά ξεκινώντας με την κυρία Καλβάλιο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε για τις παρουσιάσεις και για τον ενθουσιασμό που δείχνετε. Τρία σημεία είναι σημαντικά για το ΕΛΚ και τα οποία σίγουρα θα συμπληρωθούν από άλλους συναδέλφους. Για το Green Deal και για την καθαρή και προσιτή πράσινη τεχνολογία έχω να πω τα εξής. Βασιζόμαστε στο μελλοντικό Horizon Europe και ζητάμε τη στήριξή σας για την επαρκή χρηματοδότηση του φιλόδοξου αυτού προγράμματος για να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη ευθυγραμμίζονται και θεωρούν πως η τεχνολογία και η έρευνα αποτελούν προτεραιότητες και βέβαια ότι εκεί υπάρχει χώρος και για τον ιδιωτικό κλάδο για να έχουμε καθαρότερη και καλύτερη τεχνολογία στο μέλλον και να αποδεικνύουμε παντού πως αυτό αποτελεί Πάγει η επιδίωξή μας. Δεύτερον, η φιλοδοξία που δείχνεται στο, στο Green Deal είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει να γίνει μια σφαιρική αξιολόγηση των επιπτώσεων, γιατί δεν θα πρέπει να υποσχεθούμε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να παραδώσουμε. Και θα πρέπει να δούμε σε ποιους κλάδους μπορούμε να παραδώσουμε αποτελέσματα, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και αν έχουμε την κατάλληλη τεχνολογία. Αυτή είναι μια ερώτηση λοιπόν που έχω να σας κάνω. Το πρώτο ήταν σχόλιο. Οι επιπτωσιολογικές μελέτες έχουν προετοιμαστεί και καλύπτουν το σύνολο των φιλοδοξιών σας στους διάφορους ε, κανονισμούς που θα προτείνετε. Τέλος, για την κυκλική οικονομία, συμφωνούμε με αυτό που είπατε. Η κυκλική οικονομία χρειάζεται μια ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική και θα αποτελέσει και μια ευκαιρία. Είναι όμως πολύ λεπτή η γραμμή μεταξύ της ευκαιρίας και του βάρους για τη βιομηχανία και τις μικρομεσαίες. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν πως όντως πρόκειται για ευκαιρία και όχι ένα επιπλέον βάρος που θα οδηγήσει σε απώλεια ε, θέσεων εργασίας και δεν θα προωθήσει την ανάπτυξη αλλά θα φέρει επιβράδυνση. Ψηφιοποίηση, πράσινο πακέτο, κυκλική οικονομία, πώς θα αποτελέσουν όλα αυτά πηγή θέσεων απασχόλησης και ανάπτυξης και όχι ε, μοχλό επιβράδυνσης της οικονομίας μας. Ο κύριος Ντανίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να μιλήσω στα ρωμανικά, έτσι ώστε να κατανοήσουν και οι Ρουμάνοι ορισμένα πράγματα που είναι ενδιαφέροντος κύριε εκτελεστικό, ε, ε, είστε γνωστός ως κάποιος πολύ αποφασιστικός και όταν ε, θέσετε ένα στόχο τον υλοποιείτε. Και κανείς δεν αμφισβητεί σε αυτό το κοινοβουλίο ότι αυτό συμβαίνει. Γι' αυτό και η απόφασή μας να στηρίξουμε αυτό το New Green Deal είναι μια απόφαση που αποδεικνύεται ότι είναι κοινή ανάμεσα σε όλες τις ομάδες. Και θυμάστε, έλεγα κάτι, το New Green Deal είναι υπερβολικά σημαντικό για έναν Ευρωπαίο για να μην πετύχει. Και γι' αυτό το λόγο αυτά τα βήματα τα οποία έχετε θέσει δεν θα τα επαναλάβω, τα μοιάζονται οι περισσότεροι συνάδελφοι. Ε, ορισμένα πράγματα θα ήθελα να επιμείνω. Υπάρχουν κράτη-μέλη όπου η κατάσταση είναι εντελώ διαφορετική, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Αυτό είναι το κληροδότημα, αυτή είναι η κατάσταση. Να μιλήσω για τη Ρουμανία. Οι μελέτες που είδα, τουλάχιστον όπως παρουσιάστηκαν στο Ευρωκοινοβούλιο τον Δεκέμβριο, έλεγαν ότι η Ρουμανία θα πρέπει να, να επενδύσει 400% του ΑΕΠ της κάθε χρόνο, ξεκινώντας από φέτος, για να φτάσει του στόχους το 2030. Αυτό το πράγμα ε, δημιουργεί ερωτηματικά. Πώς μπορεί να γίνει και το πρώτο για να ε, υποδείξετε μια ομάδα όπου για αυτά τα κράτη που έχουν δυσκολίες να μπορούν να έχουν τα σχέδια έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτά τα κράτη-μελή θα μπορούσαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το 2030 και 50. Ταυτόχρονα πιστεύω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό να ζητήσουμε και για τον ελέφαντα που βρίσκεται στο δωμάτιο, διότι εδώ μιλάμε για αέριο ή μη αέριο. Ε, θα πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί αφενός ορισμένα ε, κράτη-μέλη έχουν ε, καταστάσεις για την αντακατάσταση του άνθρακα ή αλλού λένε ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι άλλο, όχι με αέριο, αλλά με κάτι άλλο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και αυτοί που είναι αντίθετοι πλαίσια αυτό το νέο Green Deal, ίσως να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και να διονύσουν αυτές τις θεωρίε που δεν, την δεν τις θέλουμε και τεχνολογίες που είναι πολύ ρηπογόνε. Γι' αυτό με απασχολεί και ε, το θέμα του πιδελταπή, γιατί... Ε, δεν καταλαβαίνω πώς θα ε, επενδυθούν ε, τα χρήματα στις ε, πρωτοβουλίες ε, του νέου Green Deal για μια νέα αποθήκευση, μια τεχνολογία που θα θα επιτρέψει ένα νέο είδος αποθήκευσης. 1% αντιπροσωπεύει τεχνολογίες αυτού του τύπου. Αναφερθήκατε στο υδρογόνο, αλλά η τεχνολογία για την παραγωγή ε, αυτή σε προσιτή τιμή και οικονομικά προσιτή ακόμη δεν είναι εκεί. Και θα πρέπει να δούμε αυτές ως προτεραιότητες και επίσης ε, στη συνέχεια στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νίκα. Και για την ομάδα Renew, ο κύριος Κριστόφ Γκρουντλέρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Καλημέρα σας. Τρεις ερωτήσεις για την ε, ψηφιακή ρήπανση, για την αφαίρεση του άνθρακα από τη βιομηχανική παραγωγή και για την διαστημική τεχνολογία στα πλαίσια του Green Deal, για το ψηφιακό. Εδώ και χρόνια το κομμάτι του ψηφιακού στην, ε, στις εκπομπές άνθρακα παγκοσμίω αυξάνεται. Αν ήταν χώρα ο ψηφιακός κόσμος θα ήταν ο πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Αν λοιπόν δεν δούμε αυτή τη διάσταση, γιατί έχουμε τα αέρια του θερμοκηπίου που ε, εκπέμπει και που θα διπλησιαστούν και θα φτάσουν στο 7,8% ε, που είναι παρόμοιο με αυτό των επιβατηγών αυτοκινήτων. Πώς θα μειώσουμε λοιπόν αυτή την ψηφιακή ρήπανση. Μήπως χρειάζονται στρατηγικά μέτρα έτσι ώστε να έχουμε μία προσπάθεια να σκεφτόμαστε περισσότερο πού εφαρμόζουμε τα ψηφιακά έτσι ώστε να προσαρμόζονται με τους κλιματικούς στόχους που έχουμε και όχι αλόγιστα να ε, ψηφιοποιούμε. Δεύτερον, για να γίνει η ευρωπαϊκή βιομηχανία σταθερή, βιώσιμη, κυκλική και χωρίς άνθρακα χρειάζονται τα εξής. Καλύτερες ενεργειακά αποδοτικές διαδικασίες και αφαίρεση του άνθρακα από τη βιομηχανική παραγωγή. Έχουμε τη βιομάζα, την ηλεκτροκίνηση, ε, το υδρογόνο, την δέσμευση άνθρακα, αλλά αυτές οι τεχνολογίες δεν είναι ακόμα επαρκώς εμπορικές. Για παράδειγμα, κύτταρα υδρογόνου. Χρειάζεται μια τεχνολογική πρόοδος που δεν έχει σημειωθεί ακόμα, με επιπλέον κόστος. Και οι βιομηχανικοί κύκλοι δεν μπορούν από μόνοι τους να προωθήσουν και να χρηματοδοτήσουν αυτή την πρόοδο. Χρειάζεται λοιπόν πολιτική που θα συνδυάζουν κανονιστικές διατάξεις και επιδοτήσει. Ποια είναι η στρατηγική σα για να επιταχυνθεί η εξάπλωση αυτών των πρακτικών που θα επιτρέψουν να μετακινηθούμε από την παραγωγή με άνθρακα. Επίσης, λίγοι πολίτες το γνωρίζουν, αλλά η διαστημική τεχνολογία έχει κομβικό ρόλο για να πετύχουμε τους κλιματικούς στόχους του Green Deal. Έγνος Κοπέρνικους Γαλιλαίο. Τα ξεχάσατε αυτά από το Green Deal. Πώς θα το αντιστρέψετε αυτό πώς θα συμπεριλάβετε καλύτερα αυτές τις διαστημικές τεχνολογίες στο Green Deal το ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γκρούντλερ, ο κύριος Μπόρκια από την ID. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζουμε κύριε Τίμερμανς και θα εκμεταλλευτώ τις άριστες γνώσεις σας των Ιταλικών και μιλάω προφανώς και εγώ Ιταλικά. Ε, κύριε Τίμερμανς, ε, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες ευαισθησίες οι οποίες έχουν προκύψει είτε σε επίπεδο κυβερνήσεων είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παραδείγματος χάρη ο Πρωθυπουργός, ο, ο Έλληνας είπε ότι η Πράσινη Συμφωνία θα φανεί πόσο δύσκολο είναι να εφαρμοστεί όταν θα αρχίσουμε να μιλάμε για την χρηματοδότησή της. Ή ο Πρωθυπουργό της Ολλανδίας είπε ότι η Πράσινη Συμφωνία είναι βιώσιμη μόνο εάν ε, υπάρχει εγγύηση και για την ε, διασφάλιση απασχόλησης. Ο Τσέχο, Πρωθυπουργό είπε ότι με την πράσινη συμφωνία δεν λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό στοιχείο. Μιλάμε λοιπόν για τρει ε, διαφορετικές ευαισθησίε, ε, οι οποίε ε, εκφράζουν και διαφορετικέ πολιτικέ ομάδε. Αυτές οι ανησυχίε δεν έχουν άμεση σχέση με πολιτικές ευαισθησίες. Και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, ο Επίτροπος Μπρετών είπε ότι ε, σε, θα χρειαστούν 25 χρόνια για να υπάρξει αυτή η μετάβαση. Ενώ ο κύριος Μπορέλ, ε, μιλώντας για τους ε, νέους ε, διαδηλωτές είπε ότι σε αυτές τις νέες γενιές ε, θα πρέπει να τους εξηγήσει κανείς ότι οφείλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους αν θέλουν να επιτύχουν αυτά για τα οποία διαδηλώνουν. Λοιπόν, αν προσπαθήσουμε να συνοψίσουμε όλες αυτές τις διαφορετικές ευαισθησίες σε σχέση με την πράσινη συμφωνία αρχίζουν να φαίνονται τα πρώτα προβλήματα. Και διερωτώ αν δεν μπορούν να βρουν τους πόρους, αν δεν μπορούν να κινητοποιήσουν ιδιωτικές επενδύσεις, είναι απαραίτητο να αναθεωρηθεί το θέμα της Πράσινης Συμφωνίας και αν ναι, τι θα σημαίνει αυτό το Συμβούλιο θα κληθεί να λάβει τις πρώτες του αποφάσεις στα πλαίσια του επόμενου Πουδουπού. Δύσκολο να επιτευχθεί η συμφωνία. Ε, τα κρατημέλη ε, δεν θα είναι ε, και πολύ πρόθυμα να συμφωνήσουν σε αυτά τα δισεκατομμύρια Τελειώνοντας, να σας πω ότι πολύ μου άρεσε αυτό που είπατε στην αρχή, ε, το δημογραφικό πρόβλημα και σε σχέση με την ε, Πράσινη Συμφωνία. Σε αυτή τη φάση, ίσως εκτός από την γενική, γενικότερη προσέγγιση, ίσως μπορείτε να μας πείτε και λιγάκι περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα. Ο κύριος Νενίστο, εκ μέρους των Πρασίνων, συντονιστής. Με ικανοποίηση διαπιστώνω πως τα εισαγωγικά σας σχόλια ξεκίνησαν με ένα κατάλογο των όσων ήδη τρέχετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το σχέδιο δράση για την κυκλική οικονομία και τα σχέδια για τα, τις βιομηχανικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολύ καλό και οι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών και να σας πω πως για την προσέγγιση της ΣΥΤΡΕ είναι προφανές πως η Ευρώπη μπορεί να λύσει το πρόβλημα του κλίματος και μπορεί να γίνει βιώσιμη αρκεί να λάβει ηγετική θέση στο χώρο της τεχνολογίας και στοχεύοντα στο να γίνει μακροπρόθεσμα βιώσιμη. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε για το πώς θα επενδύσουμε και πόσο θα επενδύσουμε. Η κλίμακα είναι τεράστια, χρειάζεται κανονιστικό πλαίσιο, τιμολόγηση, έτσι ώστε η ε, βιομηχανικοί κύκλοι να μας ακολουθήσουν, τα κακά προϊόντα να μην είναι εμπορικά βιώσιμα και βέβαια πολλές, πολλές ευρωπαϊκές επενδύσεις. Πείτε μας λοιπόν με τις ε, πι δελτα πώς πάνε τα πράγματα. Για το Horizon και για τα κλιματικά, τα επενδυτικά δεν πάμε καλά. Επίσης, τι γίνεται με την ΕΚΤ. Πώς δίνουμε τη μάχη για επενδύσεις στην πραγματική οικονομία. Τι κίνητρα θα δώσουμε. Για τα στόχου για τις μειώσεις, εμείς πρέπει να δείξουμε στον πληθυσμό μας πως έχουμε αναλάβει ηγετικό ρόλο και πριν τη Γλασκόβη να δείξουμε και στην υπόλοιπη οικουμένη πως αυτό συμβαίνει. Ποια θα είναι η πρότασή σας έτσι ώστε σε συναπόφαση να το δούμε πριν πάμε στην κόπη της Γλασκόβης για να έχουμε καλούς στόχους εν ώψη του 2030 για τις μειώσεις. Το συντομότερο δυνατόν θα ήθελα να μου πείτε πως αυτό θα συμβεί. Και σίγουρα το κοινοβούλιο εκεί θα σας στηρίξει, γιατί αυτό το 55% μείωση το στηρίζουμε ήδη εμείς. Μετά θα πρέπει να παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους κανονισμούς με την ενδυνάμωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και των στόχων εκεί, με ε, τις ΑΠΕ, με, τους ενεργειακούς, ε, με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και την ενεργειακή αναβάθμιση. Εκεί χρειάζεται αύξηση του προϋπολογισμού. Τι φαντάζεστε θα γίνει μετά την αξιολόγηση του στόχου. Τι θα προτείνετε και πώς θα πρικοδοτήσετε τα σχέδια αυτά μέχρι τον Ιούλιο του 2021, έτσι όπως μας είχατε πει στην ανακοίνωση για την Πράσινη Συμφωνία. Ο κύριος Καρασνοντέ και για την ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω και εγώ μια σειρά από ερωτήσεις. Τι προτίθεται να κάνει η Κομισιόν στο θέμα της κατανομής των προσπαθειών μείωσης. Αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Πώς θα διασφαλίσουμε τις προσπάθειες που σχετίζονται στη μείωση των εκπομπών. Το φορτίο θα πρέπει να κατανεμηθεί με διαφορετικό τρόπο μετά τον Brexit. Πώς θα γίνει η νέα κατανομή. Θα υπάρχει, ε, θα προηγηθεί μια αξιολόγηση των επιπτώσεων πριν από την απόφαση. Στο δεύτερο ερώτημα τώρα. Αυτό συσχετίζεται και με αυτό που ερώτησε ο κύριος Νίκα. Έχουμε αυτό το στόχο κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Θα συνοδεύεται και από μια αξιολόγηση του αντικτύπου ε, ε, αναλυτικά χώρα κατά χώρα. Εμείς έχουμε το ε, Ταμείο Δικές Μετάβασης, αλλά θα γίνει αποσμίση των χωρών που, μένουν, που είναι πιο πίσω από τις άλλες και αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις. Πρόσφατα, η Εθνική Τράπεζα του Βελγίου αξιολόγησε αυτό το θέμα της κλιματικής ουδετερότησης και οι αρχές της τράπεζας αποφάνθηκαν ότι η νέα πράσινη συμφωνία θα μπορούσε να είχε την ίδια επίδραση όπως η παλαιά κρίση της δεκαετίας του 70. Βέβαια ήταν απεσιόδειξη, αλλά ποια είναι η δικιά σας ε, άποψη επ' αυτού. Αυτή είναι μια προειδοποίηση από πλευράς της Βελγικής Τράπεζας. Τι πιστεύετε εσείς γι' αυτό. Άλλοι συνάδελφοι γύραν άλλα σημαντικά θέματα. Θα ήθελα και εγώ να συνεχίσω και να ε, προσθέσω με το ακόλουθο ερώτημα. Γίνεται μια συζήτηση σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία. Παράλληλα, υπάρχει και η διαδικασία του ΠΕΔΑΛΤΑΠΗ. Μήπως υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στα δύο. αν γίνουν περικοπές στις προτάσεις μας, περικοπές του προϋπολογισμού, αν μειωθεί ο προϋπολογισμός, θα υπάρχουν ε, επιπτώσεις, υπάρχει αντίκτυπος στην Πράσινη Συμφωνία που είναι τόσο φιλόδοξη ή μήπως αυτές οι δύο διαδικασίες είναι άσχετες μεταξύ τους. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Γιατί ε, όλοι αναρωτιόμαστε ποιος θα πληρώσει αυτό τα φιλόδοξα προγράμματα και σχέδια. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση και κανείς δεν... Thank you so much. Last but not least, on behalf of GUE, Madam Cornelia Ernst. Μέρους της GUE, κυρία Cornelia Ernst. Και από δική μας πλευράς ε, σας ε, συγχαίρουμε για την Πράσινη Συμφωνία, για όλους αυτές τις, τους υψηπετείς στόχους. Ε, τα πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Εγώ έχω τέσσερις ερωτήσεις. Ε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, χρειαζόμαστε ευρωπαϊκά κονδύλια που τα κράτη-μέλη κατά κάποιον τρόπο δεν θέλουν να τα καταβάλουν, προσπαθούν να βρουν με τρίκ κάποιες λύσεις. Αυτό είναι το ένα. Και κάτι άλλο που το κατέστησαν σαφές ε, και οι προναλύσανες. Πέρα από τα ενωσιακά χρειαζόμαστε και εθνικά κονδύλια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και τις, ε, την προθυμία των κρατών μελών. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να δούμε το τι θα κάνουμε καταρχήν με την ε, πολιτική λιτότητα. Αν δεν την καταργήσουμε τελείω, τουλάχιστον να τη μεταρρυθμίσουμε και να γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τον ίδιο τρόπο. Γιατί η εναλλακτική λύση είναι, αν θέλουμε, να υπάρξουν αποτελέσματα, να προωθήσουμε τις ιδιωτικοποίησεις, αλλά και αυτές βοηθάνε. Το είδαμε στην Ελλάδα. Ε, γι' αυτό λοιπόν μήπως θα πρέπει να σκεφτούμε ε, ε, να προχωρήσουμε με το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Το δεύτερο, στην Γερμανία, για τη Γερμανία θα έλεγα, είμαστε ένα έθνος του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο στη Γερμανία, ε, εντάξει μπορεί μερικοί να διαφωνείτε, αλλά το αυτοκίνητο νομίζω ότι είναι το βασικότερο σε μια οικογένεια. Εχθές λοιπόν ο κύριος Αλτμάιο, υπουργό Οικονομικών, ζήτησε και παραθέτω η αυτοκινητοβιομηχανία ε, της Γερμανίας να μην υποστεί περισσότερους και αυστηρότερους κανόνες λόγω του, της πράσινης συμφωνίας. Τέλος της παράθεσης. Εσείς τι έχετε να πείτε από αυτού, τι θα γίνει με το αυτοκίνητο, γιατί νομίζω ότι ε, δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτό, να απαλλάσσουμε την ε, αυτοκινητοβιομηχανία από την Πράσινη Συμφωνία. Κατά τα άλλα, ε, υπάρχει ένας κατάλογος ερωτήσεων που αφορά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω, η δική σας η πρόταση σχετικά με την ε, επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ποια είναι η πρότασή σας και κάτι άλλο για τον καταναλωτή. Το είπατε κι εσείς ότι θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Το πρόγραμμα είναι κοινωνικό, να ενθουσιάζει τους ανθρώπους και αν ρίξουμε λιγάκι το βλέμμα στην Ανατολική Ευρώπη, γνωρίζουμε ότι ότι η φτώχεια είναι μεγάλη και αυξάνονται και οι τιμές ενέργειας. Ας πούμε και στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε έτσι ώστε να επιτύχουμε μια κοινωνική ισορροπία και να μην αυξηθεί η ενεργειακή φτώχεια. Που τι θα σημαίνει αυτό, οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να έχουν χρήματα για να ζεσταίνονται. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν ολόκληρα σπίτια, πολυκατοικίε που δεν θερμαίνονται, κάτι που δεν επιθυμούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας δίνω το λόγο κύριε Αντιπρόεδρε για να απαντήσετε στους συντονιστές. Επτά λεπτά προτείνω για να έχουμε και περισσότερο χρόνο για τις υπόλοιπες ερωτήσεις. Το καταλαβαίνω, αλλά ελπίζω να κατανοήσουν και οι συνάδελφοι πως δεν θα μπορέσω να απαντήσω με λεπτομέρειες όλες τις ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω αμέσως. Βεβαίω η πράσινη τεχνολογία θα πρέπει να είναι οικονομικά προσιτή και όσο πιο γρήγορα αναπτυχθεί αυτή, τόσο πιο γρήγορα θα γίνει ε, αυτό. Στη βιομηχανική μας πολιτική λοιπόν και στη σχετική ανακοίνωση θα το ε, παρουσιάσουμε όπως επίσης και στο σχέδιο δράση για την κυκλική οικονομία. Δεν είστε οι μόνοι ε, που ζητήσατε την ερώτηση, που κάνατε την ερώτηση αυτή κυρία Καρβάλιο και θα σας πω πως δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τις τεχνολογίες που χρειαζόμαστε. Οι περισσότερες ήδη υπάρχουν, αλλά δεν έχουν την κλίμακα και την στήριξη που χρειάζονται για να χρησιμοποιηθούν αμέσως για να μετατρέψουν την οικονομία μας. Το πιο ενδιαφέρον είναι πως η τεχνολογία εκεί κάπου έξω βρίσκεται. Θα έλεγα δε εγώ πως βρίσκονται και τα χρήματα. Αυτό που πρέπει είναι να οργανωθούμε ως Ευρωπαίοι, να δημιουργήσουμε Ευρωπαίους πρωταθλητές σε κλάδους, έτσι ώστε να έχουμε την απαραίτητη κλίμακα, έτσι να έχουμε τις τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουμε ευρύτατα για να μεταμορφώσουμε την οικονομία μας. Γιατί? Γιατί κάποιοι αναφερθήκατε σε μια τεχνολογία η οποία είναι η πιο υποσχόμενη και έχει τόσες πολλές εφαρμογές και όπου είμαστε εμείς ε, πρωτοπόροι και όπου πρέπει να επενδύσουμε είναι το υδρογόνο. Και η οικονομία που βασίζεται στο υδρογόνο είναι μια από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες που έχει η Ευρώπη γιατί καλύπτει τόσα πολλά θέματα. Εάν μιλήσατε με τους ανθρώπους οι οποίοι στη Χαλιβουργία, για παράδειγμα στην Ευρώπη ασχολούνται, ξέρουν τις δυσκολίες. Ξέρουν πως πρέπει να αλλάξουν θεμελιωδός για να είναι βιώσιμη η χαλιβουργία και να παραμείνει στην Ευρώπη. Και οι περισσότεροι από αυτούς, αν όχι όλοι, πως το υδρογόνο είναι το κρίσιμο σημείο εδώ. Και θα συμβεί. Το ζήτημα είναι όχι το αν θα συμβεί, αλλά το αν είμαστε εμείς αρκετά δυνατοί για να το φέρουμε πέρα το συντομότερο δυνατόν για να μην έχει εξαλειφθεί από προσωπουγής μέχρι να εισάγουμε εμείς αυτή την τεχνολογία η χαλιβουργία από την Ευρώπη. Δηλαδή, κλιμάκωση με ταχύτητα για να καλύψουμε τις ανάγκες της βιομηχανίας μας. Και πιστεύω πως η χαλιβουργία αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα. Θα αναφερθώ και στην αυτοκίνητο βιομηχανία αργότερα. Στο Horizon Europe, λοιπόν, έχουμε τη δυνατότητα και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό και ελπίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στις συζητήσεις για τις PDP, πει, με συγχωρείτε, όποια θέση ευθύνη και να έχουν, είναι η αναγνώριση πως είναι φοβερά κρίσιμο να γίνει αυτή η συζήτηση γιατί μπορεί να ε, μιλήσει και να αναμίξει και να προωθήσει αλλά κυρίως να απελευθερώσει ιδιωτικού επενδυτικούς πόρους που υπάρχουν γιατί υπάρχει ενδιαφέρον για να επενδύσει κανείς αλλά θα πρέπει να υπάρχει η μακροπρόθεσμη ασφάλεια πως θα είναι αποδοτικές αυτές οι επενδύσεις και νομίζω πως αν το καταφέρουμε αυτό θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα αν το κάνουμε γρήγορα Βέβαια, θα κάνουμε και τις επιπτωσιολογικές μελέτες για οποιαδήποτε σχέδια. Και ξέρω τα τελευταία πέντε χρόνια τι σημαίνει επιπτωσιολογική μελέτη και θέλω αυτά να τα εφαρμόσω στους κλάδους στους οποίους συζητάμε τώρα και να εξασφαλίσουμε πως όσοι εμπλέκονται στους χώρους αυτούς που έχουν τη γνώση ή το ενδιαφέρον για τους κλάδους αυτούς είναι κομμάτι αυτής της επιπτωσιολογικής μελέτης που θα κάνουμε. Να αποφύγουμε σφάλματα και θυμάμαι το εξή. Τα πλαστικά μιας χρήση και την νομοθεσία η οποία πέρασε μέσα σε 8 μήνες, παγκόσμιο ρεκόρ. Γιατί καταλάβαμε πως επήγει, όχι μόνο με τους συνομοθέτες, αλλά και η κοινωνία η ίδια. Και ήταν και καλά ε, ε, προετοιμασμένοι λόγω της επιπτωσιολογικής μελέτης. Και δεν σας αποκαλύπτω μυστικά, αν σας πω πως μας στείλανε τρεις φορές να τα ξαναδούμε από την αρχή, τουλάχιστον τρεις φορές πριν υποβάλουμε τις προτάσεις μας λόγω των επιπτωσιολογικών μελετών που είχαν γίνει. Βεβαίω, πάντα ρωτά κανείς. Είναι ευκαιρία. Ποιο είναι το βάρος, αλλά αυτό το οποίο δεν απαντά κανείς σχεδόν ποτέ είναι το κόστος του να μην αναλάβουμε δράσεις. Πάντα λέμε το κόστος μιας δράσης. Και η Ευρώπη θα χρειαστεί τουλάχιστον 260 δις ευρώ επενδύσεις κάθε χρόνο για να γίνει πραγματικότητα το Green Deal. Αλλά το κόστος του να μην δράσουμε μακροπρόθεσμα ποιο θα είναι. Και αυτό θα πρέπει να το αναλύσουμε λίγο καλύτερα. Γιατί πραγματικά είναι αποκαρδιωτικό όταν κανείς ε, κοιτάξει το τι γίνεται αν δεν αναλάβει δράση, τι γίνεται με την ατμοσφαιρική ρήπανση σε περιοχές με ανθρακοριχεία. 400.000 ε, Ευρωπαίοι πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο. Για να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα της αδράνειας. Για να δούμε λοιπόν, το κόστος δράσης είναι υψηλό. Αλλά ας το αντισταθμίσουμε συγκρίνοντάς το με το εξίσου υψηλό κόστος της μη δράσης. Και αυτό χειροτερεύει ενώ καθαρότερος αέρας, καθαρότερο νερό, καλύτερες πόλεις, βιώσιμες οικονομίες βελτιώνονται εκεί. Και το λέω αυτό γιατί εγώ είμαι εγγονός ανθρακορίχου. Ρωτήστε κάποιον ανθρακορίχο και ρωτήστε αν θέλετε να γίνει ανθρακορίχος και ο γιος σας. Κάντε τους αυτή την ερώτηση και θα σας απαντήσουν μόνο αν δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα. Αν έχει άλλη δυνατότητα θα θέλανε τα παιδιά τους να κάνουν κάτι άλλο και εμείς θα πρέπει να είμαστε αυτοί οι οποίοι θα τους προσφέρουμε αυτή την ευκαιρία γιατί δεν θα συμβεί έτσι από μόνο του. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να δράσουν η Ευρώπη πρέπει να δείξει αλληλεγγύη με αυτές τις 30 περιοχές εξόρυξης άνθρακα και ανθρακοριχιών που χρειάζεται να μεταβούν και να μεταμορφωθούν σε μια άλλη εποχή. Και μας δίνει αυτό μια τεράστια δυνατότητα στον ενεργειακό μας κλάδο. Δεν μπορεί κανείς να απεμπλακεί ε, και να πει άλλο πράγμα ενέργεια και άλλο πράγμα το ψηφιακό. Αν θέλουμε τα δίκτυα να λειτουργούν, καλύτερη διανομή ενέργειας, να μην έχουμε απώλειες ενεργειακές, χρειαζόμαστε τον ψηφιακό κόσμο. Και αν χρειαζόμαστε τον ψηφιακό κόσμο, χρειαζόμαστε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, περισσότερη ενέργεια, βιώσιμη ενέργεια. Άρα λοιπόν οι ευκαιρίε είναι περισσότερε από το βάρο. Τώρα, να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση, η οποία είναι διαφορετική από κράτο μέλο σε κράτο μέλο. Δεν είναι παντού οι ίδιε οι προκλήσει. Μίλησα για περιοχέ με ανθρακοριχεία. Αν εσεί το 80% βασίζεται σε λιγνίτη, ε, είστε σε χειρότερη ε, κατάσταση παρά αν είστε ένα κράτος μέλο που χρησιμοποιείται 50% ανανεώσιμη ενέργεια. Αλλά αν δεν δουλέψουμε όλοι μαζί, αν λάβουν μέτρα μεμονωμένα τα κράτη-μέλη, οι επιπτώσεις θα είναι πολύ πιο περιορισμένες. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή την κατάσταση και πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη δεν είναι φιλανθρωπία, δεν είναι αλντρουλισμός, είναι ε, φωτισμένη ε, εγωιστική δράση. Και αυτό θα κάνει το Ταμείο για τη Δίκαια Μετάβαση και ευτυχώς στην τελευταία πρόταση του Προέδρου έχουμε φτάσει τα ε, συν 7,5 δις. Και αυτό θα μας βοηθήσει να τα καταφέρουμε. Τεχνολογία δέσμευσης και πάλι το υδρογόνο. Είμαστε στην τελευταία γενιά φωτοβολταϊκών που μπορούν να παράγουν απευθείας υδρογόνο. Αν λοιπόν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να αποθεματοποιούμε ενέργεια για αιωλική ή ηλιακή ενέργεια που θα διανέμεται μετά με σχετικά εύκολη προσαρμογή της υποδομής που έχουμε αυτή τη στιγμή για το φυσικό αέριο, έχουμε πετύχει κάτι καλό. Βεβαίως, χρησιμοποιούμε τεράστια ποσά ενέργεια σε περιοχές όπως όπως τα, ε, ε, ε, τις βάσεις δεδομένων. Ε, μας λένε η Apple και η Google, εμείς είμαστε κλιματικά ουδέτεροι. Έχουμε αυτά τα κέντρα δεδομένων που παράγουν τεράστιες ποσότητες θερμότητας και χρειάζονται για να ψυχθούν τεράστια ποσότητα ενέργειας. εντάξει, τι να τους πούμε. Αύριο λοιπόν θα λάβουμε την απόφαση για τα ψηφιακά, αλλά υπάρχει και αυτό το θέμα και θα πρέπει να το δούμε. Και θα πρέπει να κάνουμε ειλικρινές και ανοιχτέ συζητήσεις με τον ψηφιακό κλάδο και για το θέμα αυτό. Ε, οικονομία που να μην βασίζεται στην παραγωγή άνθρακα. Χρειαζόμαστε όλες τις τεχνολογίες. Εγώ εδώ για την τεχνολογία δεν είμαι καθόλου δογματικός. Ε, δεν ξέρω ε, τι θα χρησιμοποιήσουμε. Ε, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, οκ, να το κάνουμε και αυτό, να δούμε τα νούμερα, αν είναι πολύ ακριβό να το αφήσουμε, αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχω καμία ιδεολογική αντίρρηση και αυτό αλλάζει ανά κράτος μέλος. Δεν θεωρώ ότι είναι η ευφυέστερη των επενδύσεων, αλλά ας αποφασίσουν τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Και όταν ο συνάδελφος Μπρετών λέει 25 χρόνια, Κοιτάξτε, αυτό που προέρχεται από μεγάλη επιχείρηση και ξέρει πω οι επενδυτικοί κύκλοι χρειάζονται μια γενιά. Αν όμω θέλει κανεί να αναδιορθώσει έναν βιομηχανικό κλάδο, θα χρειαστεί για τη πλήρη αναδιάρθρωση ε, μια γενιά. Και γι' αυτό λέμε ορίζοντα το 2050 που είναι μια γενιά και κάτι. Για να έχουμε την ευκαιρία να πραγματικά ε, αναδιαρθρώσουμε με δύο επενδυτικού κύκλου τη βιομηχανία. Και νομίζω ότι γι' αυτό τα λέει έτσι ο Τιερή Μπρετών. Μάλιστα πρέπει να επιταχύνω. Μου έκανα νόημα. Χρειαζόμαστε να επανεκτιμήσουμε τη χρηματοδότηση του Green, Deal, του λόγω των συζητήσεων που γίνονται για σπίδα ΛΤΑΠΗ. Όχι. Αλλά θα πρέπει τις επόμενες μέρες και εβδομάδες ενδεχομένως να επιμείνουμε στο ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να δαπανίσουμε μόνο τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας για παλιές πολιτικές, να το πω έτσι πρέπει να εξασφαλίσουμε πως υπάρχει χώρος επένδυσης νέα τεχνολογία και να επενδύσουμε σε αυτά τα οποία συζητάμε. Δεν χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το ξαναδεί αυτό. Κάποια στιγμή, ναι, αλλά αυτή είναι μια εκτίμηση που γίνεται και με τις διαβουλεύσεις, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο η συμφωνία αυτή είναι κατάλληλη σε όλους τους χώρους αλλά αυτή είναι μια αξιολόγηση η οποία τρέχει, συνεχιζόμενη. Και είναι ξεκάθαρο πως χρειαστούμε μαζικές, μαζικές δημόσιες και ιδιωτικές ε, επενδύσεις σε δίκτυα, σε νέες τεχνολογίες για να συμβούν όλα αυτά. Με προκαλέσατε να μιλήσω για το δημογραφικό θέμα που αντιμετωπίζουμε ως πρόκληση. Ειλικρινά, εγώ ανησυχώ για το γεγονός ότι έχουμε τέτοια διαφορά σε κάποια κράτη-μέλη που έχουμε ερημωμένη ύπεθρο και τεράστιες πόλεις, ε, γεμάτες παράκτης περιοχές ε, και άδεια ενδοχώρα. Οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να είμαστε παραγωγικοί σε περιοχές οι οποίες είναι πιο απομακρυσμένες από ό,τι στο παρελθόν και αυτό θα απαλύνει κάπως την πίεση προς τα αστικά κέντρα αν το καταφέρομαι. Ε, έχω συναντήσει κάποιους δημάρχους τελευταίες εβδομάδες και σήμερα με τον δήμαρχο του Λονδίνου. Ναι, οι πόλεις είναι σημαντικές και θα είναι πιο σημαντικές στο μέλλον, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια συμμαχία μεταξύ υπαίθρου και πόλεων για να πετύχουμε. Και αυτή είναι μία από τις απαντήσεις στη δημοκρατική πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Το θέμα του 50-55% μείωση πρέπει να το δούμε επί τη βάση στέρεων αξιολογήσεων των επιπτώσεων και γι' αυτό δεν θα πω ποτέ, δεν έχουμε χρόνο για επιψιολογική ε, μελέτη. Και αυτό βεβαίως με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί καταλαβαίνω ότι θα θέλατε οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα να λάβουν χώρα πιο γρήγορα, όπου εκεί θα ε, παγιώσουμε το μείον 55, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μα είπαν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλύσει το κατά πόσο αυτό είναι σωστό και μπορεί να γίνει. Οπότε φοβάμαι πως αν δεν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, η στήριξη που έχουμε θα μειωθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα μας πείτε «Μα το κάνετε χωρίς να μας έχετε ε, ε, ενημερώσει και χωρίς να έχετε δει τα στοιχεία και να τα έχετε υπολογίσει». Οπότε ναι, θα γίνει η επιπτωσιολογική μελέτη και θα λάβουμε την απόφαση μόλις μπορέσουμε. Και τόσες πολλές ερωτήσεις ακόμα. Θεέ μου. Το θέμα της ουδετερότητας στις κλιματικές μέχρι το 2050 όταν λένε ότι αυτό έχει την ίδια επίδραση όπως στην πετρελαϊκή ε, κρίση, όταν λένε ότι αυτό θα οδηγήσει και στην επιτάχυνση της βιομηχανικής επανάστασης, έτσι ώστε να είμαστε πιο παραγωγικοί στο μέλλον, χωρίς αυτό το αποτύπωμα στην μητέρα γη και θα φτάσουμε στο επόμενο επίπεδο με καλύτερες θέσεις απασχόλησης πιο σύντομα, εντάξει, εάν το συγκρίνουμε με την κρίση του πετρελαίου. Αλλά αν λένε ότι η κρίση πετρελαϊκή είχε μειώσει την ανάπτυξη κλπ. κλπ. Δεν συμφωνώ. Δεν υπάρχουν τέτοιε ενδείξει ότι αυτό πρέπει να συμβεί. Θα σταματήσω εδώ και θα επανέλθω σε ορισμένα άλλα θέματα αργότερα. Και σας παρακαλώ μην αναφέρεστε στους πολίτες ως καταναλωτές. Οι πολίτες είναι κάτι παραπάνω από καταναλωτές. Καταλαβαίνουμε τι ξέρουν άμα τους βλέπουμε ως πολίτες και όχι ως καταναλωτές και τους βάζουμε σε μια ισχυρότερη θέση όταν βλέπουν τους αυτούς τους ως πολίτες και όχι καταναλωτές. Σας ευχαριστώ αυτό. Ήταν μια σειρά από ερωτήσεις. Απαντήσατε σε όλες πράγματι. Τώρα θα κάνουμε ε, δέκα σύντομες παρεμβάσεις, σύντομες ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ αυστηρό στο ένα λεπτό. Ξεκινώ με τον κύριο Μπέρνσεν ε, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, προέδρε που είστε μαζί μας ε, σήμερα το απόγευμα. Αν θέλουμε να πετύχουμε σε αυτή τη μεταβατική φάση χρειαζόμαστε και την στήριξη του υπόλοιπου κόσμου. Θα πρέπει να δώσουμε μια εμπνευστική ιστορία έτσι ώστε να καταστήσουμε σαφές τι έχουμε πετύχει. Μια από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές ε, στις βιομηχανίες μας κυρίως ε, ε, και γνωρίζω ε, στη δική σας, περιοχή, ε, δική σας περιοχή είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Είναι περιοχές που θέλουν να πάνε στην απανθρακοποίηση, αλλά χρειαζόμαστε τις σωστές υποδομές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε τις τοπικές θέσεις απασχόλησης, χωρίς να πρέπει να μεταφερθούν στις παρακτίες περιοχές. Δύο ερωτήσεις λοιπόν στην ανάλυση σας. <clears throat> Θα μπορούσατε να δείτε ε, μια προσέγγιση κατά clusters, τι clusters απαιτούνται. Δεύτερο, η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Είναι απαραίτητη. Πώς μπορούμε να τονώσουμε αυτή την τεχνολογία. Ε, θα προωθήσετε αυτό στο ρόλο σας ως εκτελεστικός ε, πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να μας οδηγήσει όχι μόνο στην ουδετερότητα του άνθρακα, αλλά και στην αηφόρο ανάπτυξη, ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, ευημερία, ευρωστία και θα πρέπει να μας βοηθήσει στο να μειώσουμε τις διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες, ελπίζω, και τις διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις κοινωνικές ανισότητες που επικρατούν. Αυτό το Ταμείο Ίσης Μετάβασης είναι εξαιρετική ιδέα, αλλά αυτή η αλλαγή θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι πραγματικά δίκαιη. Η ερώτησή μου σχετίζεται με αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω τι συγκεκριμένα μέτρα ε, θέλετε να ε, προβάλλεται έτσι ώστε να υπάρχουν πραγματικές θέσει απασχόλησης, όχι απλά επιμόρφωση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και επιμόρφωση και νεοφύης επιχείρησης, αλλά κάτι παραπάνω που θα δώσει μια όθηση στην αύξηση της απασχόλησης στις προσβεβλημένες περιοχές που το χρειάζονται. Δεύτερο, είναι η χρηματοδότηση, ε, από όσα ξέρω γίνεται μια συζήτηση στα κράτη-μέλη ανάμεσα στους καθαρούς εισφορείς και τους φίλους ε, του Ταμείου Συμμενοχής. Ε, τι στήριξη θα προέλθει από τα φρέσκα χρήματα και από το Ταμείο Συμμενοχής. Ξέρω ότι τώρα που το 50% θα πάνε μόνο σε δύο χώρε, στη Γερμανία και την Πολωνία. Ποια είναι η αποψή σα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετατροπή, αυτό το ταμείο θα χρησιμοποιηθεί με σωστό και κατάλληλο τρόπο. Ευχαριστώ κυρία Πίερ. Αξιότιμε Αντιπρόεδρε, η υποστήριξη της Πράσινης Συμφωνίας ε, μέχρι το 2050, η απομάκρυνση του άνθρακα, αυτά πράγματι μπορούν να καταστήσουν την Ευρώπη ηγέτιδα στον τομέα της τεχνολογίας. Αλλά μέχρι τώρα έχουμε αυξανόμενες τιμές ενέργειας ε, με κάποιες ε, σταθερές τιμές εκπομπών. Το ερώτημα που δείτε είναι πώς θα προχωρήσουμε. Πώς θέλετε να επενδύσετε στην έρευνα και την ανάπτυξη να διασφαλίσουμε ένα ενεργειακό μείγμα, θα επενδύσετε σε βιοσυνθετικά ε, καύσιμα, ε, οι δυνατότητες ε, από ή αν θέλετε τα δίκτυα και η αγωγή στην Ευρώπη θα είναι πιο αποτελεσματικά. Επίσης, να ρωτήσω την πρόταση του να, επεκταθεί το εμπόριο πιστοποιητικών σε όλους τους τομείς, να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια ε, για να μην, η, ε, να μην πληγούν οι ανανεώσιμες πηγές στην ενέργεια. Όλα αυτά τα στηρίζεται. Εγώ πιστεύω ότι η τεχνολογία είναι πολύ σημαντικότερη από τα, τις τιμές και το τίμημα. Ε, Βεβαίω πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ακολουθήσουμε τη στρατηγική του υπολογιστικού νεύματος αφού ε, θα ε, υπάρχουν μετακινήσεις ε, προς τα εκεί που θα έχουμε χαμηλότερες τιμές ενέργειας και στην περίπτωση αυτή δεν θα κερδίσει τίποτα το κλίμα και η πράσινη συμφωνία. Και εγώ θέλω να σας πω, είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι η Πράσινη Συμφωνία θα μετατρέψει την βιομηχανία μας, ε, τον τρόπο ζωής μας, αλλά όταν συζητάμε για αυτά τα μεγάλα θέματα, δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη λεπτομέρεια, γιατί μόνο σας το είπατε, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες, πρέπει να είμαστε συγκεκριμένοι. Δύο λοιπόν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε ε, στα απορρίμματα, στα πόβλητα, ε, στις, ε, στα πλαστικά, αλλά αναφερθήκατε και στα ηλεκτρονικά και παράγουμε πάρα πολλά, 60, 60 κιλά κατά στην Ευρώπη. Αυτή είναι η αναλογία που είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς ε, στηρίξαμε το ψήφισμα για να υπάρχει ένας ενιαίος φορτιστής για όλα τα, όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές. μπορείτε να μας ενημερώσετε λιγάκι από αυτού. Και όταν μιλάμε για απορρίμματα, ε, θα ήθελα να μπορώ να μιλήσω για τα απορρίμματα από τα τρόφιμα. Το Τούρουφ είναι ένα τρακοριχείο. Πολωνία, Τσεχία, Γερμανία εκεί, ε, ανάμεσα αυτές τις χώρες και θέλουν να το επεκτείνουν αυτό το ανθρακοριχείο. Έχετε να μας πείτε κάτι από αυτού. Ο κύριος Γκάια. Γκάια. Δεν κατάλαβα το όνομά μου, συγγνώμη. Γι' αυτό δεν πήραμε στο λόγο. Ε, αγαπητέ Φραντς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποβάλλει έγγραφα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, ε, υποβάλλει ε, νομοσχέδια. Αυτό εμένα που απασχολούν είναι η ψηφοφορία. Στις 4 Μαρτίου θα υποβληθεί ο νόμος ε, για το κλίμα και στις 10 Μαρτίου θα αναφερθεί η στρατηγική για το κλίμα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τελικά οι σκέψεις για την Πράσινη Συμφωνία, ε, πώς ακριβώς ε, μπορεί να συνδυαστεί με τη βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί αυτό που παίζει ρόλο είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε βιομηχανικά ευαίσθητες περιοχές, οι οποίες πρέπει όμως και αυτές ε, να συμβάλλουν στην ουδετερότητα των εκπομπών. Για, το, για τα νερά, τα ύδατα. Ε, ρωτώ, υπάρχουν στην Κομισιόν σκέψεις ε, σχετικά με το υδρογόνο. Επίσης, ε, υπάρχει κάποιος χάρτης πορείας για τη χρήση καθαρής ενέργειας. Ιζαμπέλα Τοβαλιέρη. Καλημέρα, Επίτροπε. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στις ε, πλαστικές ουσίες. Η Ιταλία δυστυχώς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός στην Ευρώπη και αυτό είναι ένα υλικό το οποίο υφίσταται διακριτική μεταχείριση, κυρίως από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Όσον αφορά τις πλαστικές ουσίες, είναι πολύ προχωρημένες, είναι καινοτομία και κυρίως εγγυάται την απασχόληση. 160.000 υπάλληλοι αυτοί που εργάζονται στην παραγωγή πλαστικών ε, αντικειμένων. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν πρέπει να καταδικάζουμε αυτή την παραγωγή γιατί τελικά την πληρώνουν οι εργαζόμενοι το plastic tax, ο φόρος στις πλαστικές ε, ουσίες και ύλες. Ε, αυτό κατ' ουσίαν δεν προσφέρει τίποτα παρά μόνο βλάπτει έναν κλάδο που είναι πολύ πιο βιώσιμος ε, από άλλους τομείς που δεν σέβονται το περιβάλλον. Γι' αυτό λοιπόν, παρότι είναι ρητορική η ερώτησή μου, γιατί να πρέπει να ζημιώνουμε έναν τομέα και μετά να εισάγουμε πολύ πιο ρηπογόνα προϊόντα από το εξωτερικό. Όποιο, ε, όποια ιδεολογική προσέγγιση και αν έχει κανείς σχετικά με την Πράσινη Συμφωνία υπάρχει ο κίνδυνος ε, οι δικοί μας εργαζόμενοι να μην θέλουν και να μην μπορούν να στηρίξουν ε, τέτοιου είδους πολιτικές. Κυρία Γιούτα Πάουλς. Ευχαριστώ. Το Επίτροπε. Ε, ευχαριστούμε που δεσμευτήκατε στην ε, κλινική οικονομία. Ε, νομίζω έχετε ήδη λάβει μια δυσάρεστη επιστολή από τον κύριο Altmaier, τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, όπου ο κύριος Altmaier λέει ότι για λόγους σχεδιασμού μέχρι το 2030 δεν θα, πράξει, δεν θα πρέπει να αλλάξει τίποτα στα αυτοκίνητα και Βεβαίως ε, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ε, θα έχουν χαμηλότερες εκπομπές. Εγώ θα ήθελα να ξέρω, ε, τελικά θα απαντήσει τον κύριο Αλτμαρ και αν ναι, τι θα του πείτε. Δεύτερον, είπατε ότι θα θέλατε να έχετε έναν υπολογισμό για το ποιο θα ήταν το κόστος της αδράνειας. Έχει γίνει αυτός ο υπολογισμός από το Υπουργείο περιβάλλοντος της Γερμανίας 108 ευρώ ανατόνο. Αυτή είναι η ζημιά. Με βάση τις τιμές ε, του 2016. 108 ευρώ ανατόνο, ε, Δύο δις ε, τόνοι εκπέμπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα μιλάμε για 700 τόσα δις ζημιά και αν λάβουμε την αρχική τιμή και ξεχάσουμε την έκθεση, πάμε σε 3, ε, εκατομμύρια ευρώ. Ε, και αυτά από τις δικές μας τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ο κύριος Μάρκους Πίπα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι όσον αφορά την προστασία του κλίματος και την ενεργειακή αλλαγή θα πρέπει να προχωρήσουμε. Κύριε Τίμερμανς, όμως εγώ θέλω να δω λιγάκι την ποιότητα των υποσχέσεών σας, όπως συνέβη και με την ε, στρατηγική της ε, Λισαβόνας. Ε, η ίδια είναι, γιατί μέχρι το 2050 πώς μπορείτε να είσαστε σίγουροι για την ουδετερότητα, την κλιματική. Η γεωργία, τα ζώα θα δεν μπορούμε με στα ζώα να βάλουμε ηλεκτρικό στο μάχη ε, και θα μείνουν και κάποιες άλλες ουσίες. Το ίδιο ισχύει αν θέλετε και για όλες τις καθυστερήσεις. Η Τέσλα ε, τώρα κατασκευάζει στο Βερολίνο. Οι πράσινοι διαφωνούν. Ε, χρειαζόμαστε 30 χρόνια για, μία, ε, για ένα δρόμο παράκαμψης και εσείς σε 30 χρόνια μιλάτε για κλιματική ουδετερότητα. Τα συνυπολογίσατε και τις ΜΚΟ, τις αντιδράσεις τους. Μα πώς γίνεται να έρχεστε εδώ και να μας λέτε μέχρι το 2050 θα είμαστε ουδέτεροι κλιματικά. Είναι αυτό μία υπόσχεση ή είναι αυτό μία δέσμευση. Δύο ακόμα παρεμβάσεις. Ο κύριος Τσοπισόφσκι ο πρώτος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε επανειλημμένως πει ότι το Green Deal θα αλλάξει την πραγματικότητά μας αληθεύει αυτό, αλλά ο διάβολος είναι στη λεπτομέρεια. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Σε ό,τι αφορά τις, την ιαλική ενέργεια, χρησιμοποιούμε οπτικές ίνες, η και συνθετικό πλαστικό, χρησιμοποιούμε σύνθετα υλικά. Στο παρελθόν αυτά τα συστατικά αποσυναρμολογούνταν με τρόπο που δεν ήταν φιλικός προς το περιβάλλον. Μετά το 2021 θα πρέπει να γίνει η αποσυναρμολόγηση μέχρι σε, φτάνει σε χιλιάδες τόνους ε, και στο παρελθόν όταν κλείνανε οι εγκαταστάσεις αιωλικής ενέργειας, πουλούσαμε τα εξαρτήματα στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Αφρική. Σήμερα δεν χρειάζονται και δεν θέλουν τα απορρίμματά μας. Η ερώτηση είναι η εξής. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία αυτό το ε, σχέδιο. Δεν θέλουμε να έχουμε αυτό το θέμα του κληροδοτήματος. Θα πρέπει να μάθουμε πώς να ανακυκλώνουμε και να εξαλείψουμε αυτά τα απόβλητα των εγκαταστάσεων αιωλική ενέργεια Και λίγα λόγια για το υδρογόνο. Θέλετε να διαδώσετε αυτή την τεχνολογία και είπατε ότι το ερώτημα δεν είναι ε, το ε, εάν, αλλά το πώς μπορούμε να διαδώσουμε κάτι που δεν υπάρχει. Ο κύριος Πεκαρή. Στα φιλανδικά. Arvoisa puheenjohtaja, uudet ilmastotavoitteet merkitsevät sitä, οι νέοι στόχοι του κλίματος ε, σημαίνουν ότι θα πρέπει να υπάρχουν ακόμα αυστηρότερες, περισσότερο αυστηρότερες ε, τιμές ε, στις εκπομπές για να μην έχουμε μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Η βιομηχανία καλύτερα να μην εκπέμπει δηλητηριώδη αλλά να παραμένει και ανταγωνιστική. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς ακριβώς μπορεί να ανανεωθεί η βιομηχανία έτσι ώστε οι διαδικασίες που θα εφαρμόζονται να μην ε, εκπέμπουν δηλητηριώδη αέρια και μπορείτε και να μας διασφαλίσετε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα παραμείνει ανταγωνιστική και ότι δεν θα έχουμε αντιμετωπίσει με προβλήματα λόγω της μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ε, να ξεκινήσω λέγοντας ότι πως η βάση για το Green Deal είναι η ανάγκη να μειώσουμε την αύξηση θερμοκρασίας ε, του πλανήτη κατά 0 ε, βαθμούς Κελσίου. 0,5 ε, βαθμούς Κελσίου. Διαφορετικά θα χάσουμε από τα χέρια μας τη δυνατότητα να ορίσουμε την τύχη αυτού του πλανήτη. Τώρα κάναμε κάποιες μελέτες και φτιάξαμε έναν οδικό χάρτη που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στην κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Δεν είναι απόλυτο, είναι ο δικός χάρτης. Οι επιλογές που θα κάνουμε στη διαδρομή αυτή θα αποφασίσουν αν θα πετύχουμε μέχρι το 2050. Δεν είναι εξασφαλισμένο, εξαρτάται από τις επιλογές μας. Αλλά οι επιλογές που έχουμε στον οδικό χάρτη μπορεί να μας οδηγήσουν στο να είμαστε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος μέχρι τότε είναι πιεστική ανάγκη αυτή σε επίπεδο κοινωνιών και πιστεύω πως ο πλανήτης μας θα μας θυμίζει κάθε χρόνο πως χρειάζεται κάτι τέτοιο. Το βλέπουμε καθημερινά πια. Και πιστεύω πως έχουμε πραγματικά μια ευκαιρία γιατί μπορούμε να το συνδυάσουμε με την βιομηχανική επανάσταση η οποία θα μας φέρει σε μια νέα οικονομία, με νέες θέσεις εργασίας. Είμαι πεπισμένο πως γίνεται. Θα είναι εύκολο. Μα τι λέτε, καθόλου εύκολο, πάρα πολύ περίπλοκο. Αλλά Πόσο διασκεδαστικό είναι να κάνει τα πράγματα κανείς που είναι εύκολα. Αλλά έχουμε να αφήσουμε ένα πλανήτη και μία ήπειρο στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας που θα έχει κάποιες πιθανότητες επιβίωσης που θα βασίζεται στις δικές μας καινοταμίε δυνατότητες και ιδέες για να αλλάξει. Δεν είναι η στρατιωτική, η στρατιωτική ισχύς που θα μας κάνει ε, πρώτους στον κόσμο. Δεν είναι ο αριθμός Ευρωπαίων που θα μας κάνει πρώτους στον κόσμο. Είναι οι, πώς, οι ελκυστικές μας κοινωνίες που θα μας κάνουν πρώτος στον κόσμο και αυτό θα μας το παραδώσει το Green Deal. Και βέβαια θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία των clusters. Δηλαδή, θα μιλήσουμε σε γενικές γραμμές για το τι θέλουμε να πετύχουμε και μετά θα ομαδοποιούμε ανακλάδο. Τι σημαίνει αυτό για κάθε κλάδο. Δηλαδή χημική βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, χαλιβουργία, ε, γεωργία κτλ. Έχουν κοινά στοιχεία, αλλά έχουν και ιδιάζοντα χαρακτηριστικά και προκλήσεις που χρειάζονται συγκεκριμένη προσέγγιση. Ένας από τους κλάδους που δεν αναφέραμε ακόμα και θέλω να αναφέρω εδώ, γιατί είναι μια από τις μεγαλύτερες ε, ευκαιρίες που παρουσιάζεται στην κοινωνία μας, είναι το 80% των κτηρίων που θα έχουμε το 2050 ήδη είναι έτοιμα. Και τα κτίρια αυτά χρειάζεται να προσαρμοστούν, να μονοθούν, να γίνουν κλιματικά ουδέτερα, να αλλάξουν χρήση ενέργειας. Είναι η μεγαλύτερη δυνατότητα δημιουργία θέσεων εργασία που υπάρχει και μπορούμε να τα κάνουμε. Τα κεφάλαια υπάρχουν. Μιλήστε στι τράπεζε, στην ΕΤΕΠ, είναι επενδύσεις χωρίς κίνδυνο ουσιαστικά και μπορεί να γίνει. Είναι θέσεις εργασίας, τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε από την Ευρώπη, θα πρέπει να γίνουν εδώ. Ακόμα και η ανακύκλωση των παλιών ε, ανεμογεννητριών, για παράδειγμα. Μπορούμε να το κάνουμε στην Ευρώπη. Εδώ. Πιστεύω δε, και αυτό είναι ένα σχόλιο για τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα, Χρειάζεται εκεί να κάνουμε κάποιες ε, προσπάθειες. Τεχνικά γίνεται, αλλά εξαρτάται με το που είσαι. Αν είσαι στην παραλία είναι εντάξει. Αν είσαι στην ενδοχώρα πολύ πιο δύσκολο. Έχουμε όμως ευκαιρίες για κάποιου κλάδους και κάποιες περιοχέ, ε, περιοχές, αλλά δεν είναι και το μαγικό ραβδί που θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά σε μια μεταβατική περίοδο μπορεί να είναι τεράστια η σημασία του και η αξία του. βεβαίω θα πρέπει να δούμε και τα συγκεκριμένα μέτρα στο Ταμείο για τη Δίκαιη Μετάβαση και είμαι πεπισμένος πως δεν θα τα καταφέρουμε εάν οι πολίτες μας δεν πιστέψουν πως είναι για το καλό τους. Αν δεν αποτελέσουν τμήμα της προσπάθειας. Εάν θελήσουν να κάνουν θυσίες γιατί γνωρίζουν πως θα κερδίσουν κάτι αυτοί και τα παιδιά τους, εντάξει, αλλά αν δούνε μόνο που ζητάμε θυσίες, δεν θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε. Οπότε το Ταμείο αυτό θα πρέπει να το λάβει τούτο υπόψη. Για την ενέργεια πρέπει να το δούμε. Δίκτυα, πιέζει, εγκαταστάσεις αποθεμάτωσης, όχι μόνο μπαταρίες, αλλά το υδρογόνο θα αποτελέσει ε, ένας από μία από τις μεγαλύτερες δυνατότητες αποθεματόπισης αποθεματοποίηση ενέργειας. Ενεργειακή φορολόγηση. Το σύστημα σήμερα βασίζεται στα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να αλλάξει. Ένα πιο πράσινο σχέδιο φορολόγησης. Διστάζουν τα κρατημέλη να το συζητήσουμε, αλλά είναι αναπόφευκτο. Σε αρκετά κρατημέλη ενέργεια επιδοτείται παρόλο που προέρχεται από ορυκτά καύσιμα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα σταματήστε τι επιδοτήσεις και περάστε σε άλλη μορφή ενέργειας και τριπλασιάζουμε και του λογαριασμού σας. Ε, δεν γίνεται αυτό. Ηλεκτρονικά απόβλητα. Τεράστια πρόκληση. Ανακύκλωση. Είδα την απόφαση για, την, για τον ενίο φορτιστή. Είναι κομμάτι του πακέτου κυκλικής οικονομίας. Όχι μόνο οι φορτιστές και τα καλώδια και η βιωσιμότητα των καλωδίων. Ανθρακοριχεία στην Πολωνία. Θα τα πω με την πολωνική κυβέρνηση αυτή την εβδομάδα για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Να είμαι κι εγώ πιο ενημέρος. Πλαστικά. Εμείς αφαιρέσαμε 10 πλαστικά μιας χρήσης για τα οποία έχουμε βιώσιμες εναλλακτικέ που δεν δημιουργούν πρόβλημα στον καταναλωτή. Αλλά όταν φύγουν αυτά τα 10 πιο δημοφιλή πλαστικά μιας χρήσης, ε, ουσιαστικά αφαιρείς το 70% που μπαίνουν στους ωκεανούς μετά και στα ποτάμια και στα νερά. Είναι καταπληκτικό πριν το πλαστικό. Καταπληκτικό. Και το χρειαζόμαστε γιατί η βιωσιμότητα είναι πιο μακρά διάρκεια, πιο δυνατά, πιο ελαφριά τα προϊόντα, αλλά είναι και επικίνδυνο. Τα, πλαστικά μια χρήση και τα μικροπλαστικά είναι επικίνδυνα για την υγεία μα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αν ήμουν από την Ιταλία, δεν θα ήμουν τόσο απόλυτη στην υπεράσπιση των πλαστικών. Πηγαίνετε να ρίξετε μια ματιά και στα νερά και στι παραλίε στην Ιταλία που είναι ε, μαργαριτάρι της ε, ε, Ιταλικής οικονομίας, ο τουρισμός, θα καταστραφεί αν δεν βγάλετε από το περιβάλλον τα πλαστικά. Δεν έχω τίποτα εναντίον των πλαστικών, αν είναι βιώσιμα. Τα χρειαζόμαστε, αλλά όχι τα μίας χρήσης. Να πω κάτι για την αυτοκινητοβιομηχανία, γιατί ακούστηκε η επιστολή. Θα κάνουμε και τη μελέτη επιπτώσεων και θα δούμε τα επόμενα χρόνια αν θα είχαμε πλέον νομοθεσία. Ο κλάδος αντιμετωπίζει τεράστια πρόκληση και για πρώτη φορά φέτος είμαι πεπισμένος πως έλαβε το μήνυμα και θέλει πια να κάνει τις απαραίτητες αλλαγές. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στα περισσότερα κράτη-μέλη αυτές οι αλλαγές έχουν τεράστιους κινδύνους για την απασχόληση. Αυτό αποτελεί ανατροπή σε ένα μεγάλο κλάδο της βιομηχανικής Ευρώπης. Πρέπει να γίνει και όσο το δυνατόν νωρίτερα καλύτερα. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως θα δώσουμε ευκαιρίες σε όσους εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία για να συνεχίσουν εκεί σε άλλες θέσεις, με άλλες δεξιότητες ενδεχομένως ή να πάνε σε άλλο κλάδο που θα χρειάζεται κόσμο σύντομα. Το μήνυμα λοιπόν είναι ότι η αυτοκινητομηχανία στην βιομηχανία στην Ευρώπη καταλαβαίνει πως θα πρέπει να φύγει από το κινητήρα εσωτερικής καύσης, χρειάζεται μαζικές επενδύσεις και χρειάζεται να συνεργαστεί μαζί μας. Αλλά και εμείς πρέπει να καταλάβουμε πως είναι τόσο τεράστια αυτή η μεταμόρφωση πως δεν θα πρέπει να χαθούν θέσεις εργασίας χωρίς λόγο και να προσφέρουμε νέες θέσεις σε αυτούς που τις χρειάζονται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, όταν μιλήσει κανείς ε, και για φορτηγά και άλλα οχήματα, το πράγμα δυσκολεύει. Έχουμε ακόμα τέσσερις ε, παρεμβάσεις και πρέπει να απαντήσετε και να έχουμε και τα τελικά συμπεράσματα, αλλά έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Ο κύριος Κόμπουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. κύριε Αντιπρόεδρε, συμφωνούμε όλοι ότι η περιοχή Σαλίζια ε, που έχει ανθρακοριχεία αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Χρειάζονται σοφές και σωστέ αποφάσει και σωστά μέτρα. Έχω μία ερώτηση που αφορά ε, στο εξή. Ακούσαμε χθε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι δύο δις ευρώ προβλέπονται για την Πολωνία για το Ταμείο ε, Δίκαιη μετάβαση. αλλά μπορεί να πάρει τα μισά αν δεν έχει πετύχει μέχρι το 2050 η Πολωνία την κλιματική ουδέτερη η Κομισιόν τι πιστεύει γι' αυτό και δεύτερον πρόσφατα αναφέρθηκε στην Επιτροπή των Περιφερειών από την Ένωση Πολωνικών, σε Ένωση Πόλεων ότι ε, κονδύλια θα δοθούν και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εσείς τι πιστεύετε για όλα αυτά, Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια φιλοσοφική ερώτηση που αφορά στην ε, κλιματική αλλαγή. Τι πρέπει να πετύχουμε το 2050, κλιματικά ουδέτερη οικονομία ή ε, ουδέτερη ε, ατμόσφαιρα. Η κλιματική αλλαγή είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση και εμείς εστιάζουμε την προσοχή μας στην μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Τι είναι λοιπόν η κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Επίσης, ένα άλλο εξίσου σημαντικό ε, στοιχείο για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή είναι οι αρνητικές εκπομπές. Αυτό δεν έχει σχέση με την δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα. Αυτές όμως οι αρνητικές εκπομπές πολλές φορές αγνοούνται. Αν δείτε τι σημαίνει στην τεχνολογία, στην βιτεχνολογία, θα δείτε ότι εκεί υπάρχουν ελπιδοφόρες εξελίξεις αυτή θα μπορούσε να είναι μια ρηξικέλευτη τεχνολογία, η δική μου ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί η Επιτροπή δεν αρχίζει να εξετάζει νέες τεχνολογίες και τις αρνητικές εκπομπές ε, που θα μπορούν να είναι πολύ ε, χρήσιμο. Κύριε Πρόεδρε, η επιτυχία του, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ε, συνδέεται με προϋποθέσεις, με τις εξής. Πρώτον, πρέπει να διασφαλίσουμε να είναι δίκαιη η μετάβαση. Οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να έχουν μία συμφωνία όπου το μεγαλύτερο τμήμα του βάρους ε, ε, αφορά και μετακυλείται σε εκείνους που είναι όμως ε, οι υπέτειοι. Το δεύτερο, ε, για μας είναι απαράδεκτο να μην υιοθετηθεί η ευρωπαϊκή πρόταση. Να μην εποφεληθούν οι πολίτες και να μην εφαρμόζονται προτάσεις χωρίς αποκλεισμούς. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι χρειαζόμαστε νέες δυνατότητες χρηματοδότησης, νέα κεφάλαια. Η Κομισιόν πώς προτίθεται να διασφαλίσει αυτήν την δίκαιη μετάβαση χωρίς να αφαιρέσει κονδύλια από άλλους ε, τομείς. Κονσάλες Καστάντες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ κύριε Τίμερμανς. Ε, θα συνεχίσω στα Ισπανικά. Ε, μιλήσατε για την ε, Πράσινη Συμφωνία. Έχουμε ε, προτάσεις για το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο είναι δυνατόν να βελτιωθούν τα κριτήρια να συμπεριληφθεί ενδεχομένως και η ανεργία. Στην Γαλλική, παραδείγματος χάρη, θα κλείσουν οργία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, καταβάλλετε προσπάθειες ε, για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Όταν ε, θα έχουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία σύζευξη θεμάτων και να μπορέσουμε τελικά να έχουμε παντού ενέργεια. Αυτός ο πέμπτος κατάλογος Μήπως θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε για την ε, παραγωγή ενέργειας. Τι είδου δυνατότητες υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε ε, Τινμάνς είπατε ότι οι πολίτες ε, πρέπει να προσπαθήσουν ε, να εκμεταλλευτούν ε, την Πράσινη Συμφωνία και μετά ε, παραπέμψατε στα χρήματα φορολογουμένων. Υπάρχει λοιπόν αυτή, αυτός ο παραμβατικός χαρακτήρας. Βλέπω ότι γελάτε, χαμογελάτε, αλλά και εγώ τα βρίσκω όλα αυτά χαριτωμένα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω ένα άλλο ερώτημα που αφορά τον κορονοϊό και τη βιομηχανία μας. Γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε μία φάση αποβιομηχάνηση τα τελευταία χρόνια από τον Νοέμβρη μέχρι το Δεκέμβρη του 2019 μειώθηκε η βιομηχανική παραγωγή κατά 2,1% και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί μάντες παραγωγής ε, δεν λειτουργούν στις ε, βιομηχανίες γιατί λείπουν οι πρώτες ύλε που είναι απαραίτητε για παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές σε μεγάλο βαθμό ερχόντουσαν από την Κίνα και λείπουν. Στο μέλλον πώς θα μπορέσετε να διασφαλίσετε τον εφοδιασμό αν θέλουμε να παράγουμε εδώ στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο περισσότερα δευτερογενή προϊόντα. Κυρία Μαρή Τουσάν, έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω κι εγώ στη μητρική μου γλώσσα. Κύριε Τίμερμαντ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω να μιλάτε για τον πλανήτη Γη, για τους απαραίτητα ηλεκτρικά δίκτυα, για την εγκατάσταση των ορυκτών καυσίμων. Σας χαίρομαι όταν σας ακούω να μιλάτε για το υδρογόνο ΑΠΕ, αλλά θα ήθελα να επανέλθω και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σα σε αυτή την ε, λίστα. Ε, είπατε μέσω Twitter ότι για να πάρουμε χρηματοδότηση από την ΕΕ θα βρίσκονται, τα προγράμματα θα πρέπει να στηρίζουν την φιλοδοξία μας για το Green Deal. Θα ήθελα να μας, εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Για να ελοπίσετε το Green Deal, συμφωνείτε ότι το φυσικό αέριο δεν μπορεί πια να αναπτυχθεί, δεν μπορούμε να έχουμε άλλες εκμεταλλεύσεις. Τι ε, θα κάνετε για να αξιολογήσετε τα έργα που υπάρχουν στο κατάλογο αυτό αυτή τη στιγμή. Θα λάβετε υπόψη την ε, ύπαρξη της ΑΣΕΡ και άλλες μελέτες που έγιναν και δημοσιεύθηκαν ε, λίγες μέρες πριν από την τελική οριστικοποίηση αυτού του καταλόγου που θα κάνετε ε, μελέτες εξερώχησης των επιπτώσεων, ε, σκοπιμότητας. Ε, εάν θέλετε να δώσετε κάποια συγκεκριμένη απάντηση, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κοντούρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία μέσω του μηχανισμού δίκαιης μετάβασης προβλέπει τη στήριξη των περιφερειών που βασίζονται στην παραγωγή άνθρακα και λιγνίτη και έχουν δεσμευτεί για κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Για να προχωρήσουμε όμως σε μια δίκαιη μετάβαση για τις τοπικές κοινωνίες θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καταρτήσουν κοινωνικά δίκαια και υλοποιήσιμα σχέδια απολιγνητοποίησης. Στη χώρα μου, στην Ελλάδα, μετά από την απόφαση της κυβέρνησης για απολιγνητοποίηση με ασφικτικό deadline μέχρι το 2023, η Δυτική Μακεδονία και η Μεγαλόπολη βρίσκονται ενώπιον του κινδύνου κοινωνικής κατάρρευσης. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως υποστηρίζουμε την απολιγνητοποίηση, όμως η απόφαση αυτή λήφθηκε χωρίς το σχέδιο της κυβέρνησης να μπορεί να εξασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και τη βιωσιμότητα της μετάβασης και χωρίς να υπολογίζει το αρνητικό αντίκτυπο που θα έχει στις τοπικές κοινωνίες. Σας ερωτώ λοιπόν πώς η Επιτροπή σχεδιάζει να υποστηρίξει ουσιαστικά τις περιφέρειες αυτές καθώς το ποσό των 293 εκατομμυρίων ευρώ που τους ανολογεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης δεν επαρκεί για να επιτευχθεί μια κοινωνικά δίκαιη και όχι βίαιη μετάβαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, uh,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 θέμα είναι ότι έχουμε πάρα πολλές ε, ανεμογεννήτριες σε σχέση πάντα με την νεολική ενέργεια, η οποία σε 20 χρόνια, οι οποίες θα πρέπει ε, να αντικατασταθούν. Εν τω μεταξύ με οι ανεμογεννήτριες ε, ε, σκοτώνουν πάρα πολλά ζώα και πάρα πολλά πουλιά. Ε, εξάλλου, το τι παράγεται από ενέργεια, αυτό το κοιτά κανεί πάντα αποκομμένα. Θα πρέπει όμως να συνυπολογιστούν και άλλοι παράγοντες, γιατί η ολική ενέργεια, κατά την άποψή μου, δεν είναι επουδενή ιδανική. Η ενέργεια και το ρεύμα έχει και αυτό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 Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια σε εσά την τελευταία μιλήτρια που ήταν τόσο γρήγοροι. Δεν ξεπεράσει το χρόνο σας. Συγκεκριμένε τώρα απαντήσει σχετικά με την Πολωνία. Νομίζω ότι η φιλοδοξία μου είναι να διασφαλίσω ότι η Πολωνία θα δεσμευτεί και αυτή για τους ε, στόχους του 2050. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό για όλου μα να δεσμευτούν όλα τα κράτη-μέλη και μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο ε, μέσα από το Ταμείο τη δική μετάβαση και άλλα μέτρα που θα λάβουμε, μπορούμε να αποδείξουμε ότι όλα αυτά είναι εφικτά. Βεβαίω και θα συνεργαστούμε και άμεσα με την τοπική αυτοδιοίκηση κατά τα επόμενα έτη. Έχω συζητήσει με του Δημάρχου, έχω συζητήσει με ήδη υπάρχουσε δομέ, όπω η Επιτροπή των Περιφερειών ή το C40 ή άλλε πρωτοβουλίε, ε, τι Ενώσης των δημάρχων. Ε, θα δουλέψουμε με κεντρική κυβερνήσει, αλλά και συμπληρωματικά τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί ποικίλουν πάρα πολύ οι συνθήκε τη τοπική κοινωνία και μέσα στο ίδιο κράτο μέλο. Και επιπλέον, ε, αν το κάνουμε αυτό, οι άνθρωποι θα ε, δείξουν μεγαλύτερο ενθουσιασμό και μεγαλύτερη στράτευση. Ε, κοιτάξτε, και καθαρά πρακτικά. Η συζήτηση δεν είναι μόνο φιλοσοφική, είναι και πρακτική. Το κατά πόσον θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα. Ε, είναι πολύ σημαντικό βέβαια να έχουμε μια τέτοια οικονομία, όχι ουδέτερη κοινωνικά, ουδέτερη προς το κλίμα. Οι πολίτες μας λένε ότι θέλουμε καλύτερη ποιότητα του ατμόσφαιρα. Ε, και δεν θα δεχτούμε πια το οικονομικό επιχείρημα ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά ε, για να υπάρχουν θέσει απασχόλησης. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι θέλουν πιο πράσινες πόλεις, ε, θέλουν πιο πράσινες περιφέρειες. Οι άνθρωποι θέλουν να σταματήσουν αυτό που ο Μακρόν αποκάλυψε «εκοσίδ». Ε, δεν θέλουν να εξαφανιστούν ε, πολλά είδη ε, του ζωικού βασιλείου. Οι άνθρωποι θέλουν πιο καθαρό νερό. Δεν πρόκειται μόνο για την απολιγνητοποίηση και την αφαίρεση του άνθρακα από την οικονομία μας. Οι άνθρωποι θέλουν μια καλύτερη ζωή, βιώσιμη ζωή. Υπάρχει βέβαια και άλλη πλευρά του νομίσματος που βεβαίως αυτό σημαίνει δεν λέμε ότι δεν θα υπάρχουν πια καθόλου εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Λέμε ότι η ε, μητέρα γη ε, δεν πρέπει να της δημιουργήσουμε αναταραχή και εσείς ε, πολύ σωστά λέτε και αν αντεπιχειρηματολογείτε ότι χρειαζόμαστε χώρους όπου να υπάρχει περιτόριο για την απορρόφηση του άνθρακα. Πολύ σωστά λέτε ότι πρέπει να υπάρξουν τεχνολογίες εξελίξεις στο θαλάσσιο περιβάλλον, στα φύκια, την εκμετάλλευσή τους, στα δάση, αναδάσωση. Γιατί? Για να έχουμε καλύτερη δέσμευση του άνθρακα, να κάνουμε κάτι καλύτερο στη βιοπικιλότητα. Δεν είναι απλά και μόνο το να αφαιρεθεί ο άνθρακα από την οικονομία μα. Το θέμα είναι πώ θα επαναφέρουμε μια ισορροπία στην ανθρωπότητα, πώ θα συμβιώνει καλύτερη η ανθρωπότητα με το περιβάλλον. Γιατί μερικέ φορέ λέμε ότι να σώσουμε τον πλανήτη. Μα δεν πρέπει. Κανεί δεν είπε να σωθεί ο πλανήτη. Μόνο θα φέρνει ο πλανήτη μια χαρά μόνο του και με εμά και έχοντα ξεφορτωθεί εμά. δεν είναι να σώσουμε τον πλανήτη, την ανθρωπότητα να σώσουμε. Να έχουμε ένα πλανήτη όπου οι άνθρωποι να ζουν καλά. Είμαστε 10 δις. Ε, να ζούμε με έναν τρόπο που να είναι πιο δίκαιο, Να λαμβάνουμε υπόψη μα τις φιλοδοξίε και άλλων ανθρώπων υπανάπτυκτων σε άλλα μέρη του κόσμου που θέλουν και εκείνοι να ζουν όπω και εμεί. Αυτό είναι σημαντικό να το έχουμε κατά νου και ξεφεύγει από τα καθαρά οικονομικά. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι ένας από εκείνους που λέει όλα αυτά είναι εύκολα, ότι ε, δεν θα έχουμε καμία απογοήτευση, ότι δεν θα σκοντάψουμε. Όλα αυτά θα γίνουν όπως συμβαίνει πάντα. Όμως ε, το σημείο κίνησης θα πρέπει να είναι ότι δεν είναι ότι είναι μόνο το σωστό πρέπει να γίνει, γιατί συγγνώμη αλλά είναι, αυτό είναι και εφικτό, γιατί συγγνώμη είναι εφικτό. Και όλοι πρέπει να πιστούμε για κάτι τέτοιο, ακόμα και αν απογοητευόμαστε μερικές φορές. Παρ' αυτά ε, ξεπερνάμε την απογοήτευση και συνεχίζουμε. Και μερικές φορές ε, το βρίσκω παράδοξο το ότι ορισμένα κόμματα που ε, κατακρίνουν την κρατική παρέμβαση είναι τα ίδια κόμματα που σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούν την κρατική παρέμβαση για να περικοπούν οι αστικές ελευθερίες. Τέλος πάντων, το είπα και αυτό, απλά ήθελα να το πω. Ε, αυτά βέβαια μας οδηγούν στο να αναζητάμε κονδύλια και πέρα από τα κρατικά κονδύλια για να γίνουν επενδύσεις. Η εντύπωσή μου τους τελευταίους μήνες είναι ότι πάρα πολλοί ε, οικονομικοί παράγοντες και επενδυτές απελπισμένα ψάχνουν να βρουν καλές επενδύσεις. Αν λοιπόν όλα αυτά είναι αξιόπιστα και αν εμείς είμαστε εκείνοι που προσφέρουμε ε, το περιβάλλον για την ε, προβλεψιμότητα και τη σταθερότητα, τότε νομίζω ότι έτσι μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις. Και αυτή είναι και η απάντηση ε, στο πού θα ε, φτάσουμε. Αν μιλήσει κανείς ε, με ανθρώπους που θέλουν να κάνουν περισσότερα πράγματα σε αυτόν τον τομέα, πολύ συχνά λένε αν πάω στις Ηνωμένε Πολιτείε, παίρνω άδεια μέσα σε μια εβδομάδα και αυτή ε, ε, έχει αξίε ολόκληρη την Αμερική, για ε, επενδύσεις μιλάμε, στην Ευρώπη λένε χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο καιρό. Ναι, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι στην Ευρώπη έχουμε πάρα πολλές νοηθείς επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν προχωράνε. Και γι' αυτό να κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Σίγουρα η επιρροή μας είναι περιορισμένη, αλλά αυτή ε, θα πρέπει ε, να είναι σωστή επιρροή και ε, στη γραφειοκρατία μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μερικοί από εσάς ίσως περιμένετε μία απάντηση για τον κατάλογο PCI, για πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος. Να σας πω ότι αυτό αυτό, σε αυτό έχουμε δεσμευτεί. Νομίζω το Κοινοβούλιο έλαβε τη σωστή απόφαση, αλλά θέλω επίσης να πω με απόλυτη σαφήνεια ότι η απόφαση αυτή θα είναι συνάρτηση του ότι δεν θα επενδυθούν ε, σε τομείς που, όπου θα χαθούν τα χρήματα. Βεβαίως, ορισμένοι από εσά θέλετε να ξέρετε ακριβώ ε, το τι και πώς και πώς. Εντάξει, το καταλαβαίνω, δουλειά σας είναι, αλλά τι να κάνω και εγώ. Δική μου δουλειά είναι σήμερα να σας πω ότι σας το υπόλοιπα υπόσχομαι και μετά από λίγο καιρό να με τσεκάρετε, να με ελέγξετε και να δείτε αν θα τα έχω τηρήσει όλα αυτά ή όχι. Ε, έτσι παίζει το παιχνίδι. Ε, έτσι θα προχωρήσουμε. Ε, σε αυτή τη φάση μόνο αυτό μπορώ να πω. Όσον αφορά τώρα την Ελλάδα, κοιτάξτε, νομίζω πρέπει να τα ξαναπούμε, να επανέλθω. Γνωρίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι θετική ε, απέναντι σε αυτά που κάνουμε. Ξέρω ότι υπάρχουν προβλήματα σε κάποιες περιοχές, όμως να πω και κάτι γενικότερο. Θα πρέπει να επαναπροσανατολίσουμε τα υπάρχοντα κονδύλια, δηλαδή δεν είναι μόνο τα επιπλέον, είναι και αυτά που υπάρχουν ήδη στο Ταμείο Συνοχή, στα διαρθρωτικά ταμεία, στην κοινή γεωργική πολιτική, να αναπροσανατολίσουμε τα κονδύλια που έχουμε, έτσι ώστε ό,τι κάνουμε να μας οδηγεί στη σωστή κατεύθυνση. Και ε, ξεκινάμε με το 25%, λίγο αυτό, και μετά θα προχωρήσουμε σε υψηλότερο επίπεδο. Ε, τελευταία μου τώρα παρατήρηση, για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, γιατί ετέθη και αυτό το ερώτημα. Ε, κοιτάξτε, εγώ δεν έχω καμία δέσμευση απέναντι στην πυρηνική ενέργεια. Και ξέρουμε ότι από την πυρηνική ενέργεια δεν προκύπτουν εκπομπές, αλλά προκύπτουν άλλα προβλήματα, πυρηνικά απόβλητα και συναφή. Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σέβομαι τα κράτη-μέλη ε, που έχουν τη στάση ναι ή όχι για την πυρηνική ενέργεια. Εμείς ε, δεν θα παρέμβουμε στα κράτη-μέλη. Το μόνο που λέω είναι να Κοιτάξτε λίγο τους αριθμούς. Αυτή η επένδυση είναι ευφύης επένδυση και για μένα, κοιτάγοντας τους αριθμούς, το συμπέρασμά μου είναι ότι είναι πολύ πιο ευφυές το να επενδύσει κανείς σε βιώσιμες ε, εγκαταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε επίπεδο αρχή δεν έχει καμία αντίρρηση απέναντι στην ποινική, ε, ενέργεια. Εγώ σα λέω, δέστε μόνο του αριθμού. Και οι αριθμοί απλά δείχνουν μία αύξηση. Δέστε λιγάκι τι γίνεται στη Γαλλία. Ε, η Γαλλία που είναι μεγάλος οπαδός της πυρηνικής ενέργειας και αυτοί ε, αναπροσανατολίζονται προς βιώσιμη ενέργεια και ξέρετε γιατί, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει αύξηση. Αυτό το δείχνουν οι αριθμοί. Και βεβαίως ε, ε, η βιώσιμη ενέργεια έχει προβλήματα. Βεβαίως ε, πρέπει να διασφαλίσουμε η βιώσιμη ενέργεια να γίνει πιο αξιόπιστη στο μέλλον. Αλλά αυτά είναι ένα κομμάτι της μετάβασης και μπορούμε να το πετύχουμε όλο αυτό με τη δική σας τη βοήθεια. Thank you very much. Uh, thank you very uh, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Η κατεύθυνση λοιπόν είναι σαφής. Ε, πολλοί από τους συναδέλφους μου θα μιλούσαν για κατεπίγουσα ανάγκη. Ε, πράγματι συμφωνούμε όλοι ότι κάτι πρέπει να γίνει. Διχασμένοι είμαστε στο πώς μπορούμε να τα πετύχουμε όλα αυτά. Ξακολουθούμε να συζητάμε για την πυρηνική ενέργεια και ε, πολλοί διερωτώνται πώς η δίκαιη μετάβαση μπορεί να είναι αποτελεσματική. Αλλά είμαστε ευγνώμονες που ήρθατε σήμερα κοντά μας και με μεγάλη μας χαρά να συνεχίσουμε το διάλογο και να συζητήσουμε για το πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. Ε, παρακαλώ να βγείτε από την αίθουσα εκτός από τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε και τη Γραμματεία και τους βοηθούς για να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση κυκλισμένων των θυρών σε τρία λεπτά. Σας ευχαριστώ.